Bien. <coughs> Oh, oh, Ça sonne un peu creux, mais bon. Καλησπέρα. Δεν είμαστε και πολλοί. Je pense que 5 minutes, c'est bien. Hein? On va pas pénaliser euh, les bons élèves. Λοιπόν, Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν νομίζω να υπήρξαν αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη. Την εγκρίνουμε λοιπόν. Δεν έχω ειδικέ ανακοινώσει ω πρόεδρο. Ή μάλλον ο κανονικό πρόεδρο ζητεί συγγνώμη που είχε ανελειμμένε υποχρεώσει και δεν βαρίσταται. Πάμε στο πρώτο σημείο τη σημερινή διάταξη. Να εξετάσουμε την πρώτη του τροποποιεί την οδηγία τη σχετική με τη διαχείριση τη ασφαλεία των οδικών υποδομών. Στην κυρία Αγιούτο θα δώσουμε το λόγο να μας παρουσιάσει την πρόταση. Κυρία Συγήτρια, έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Δυστυχώς Δευτέρα απόγευμα, ξέρεις, συνεδριάσεις δεν είναι και περισσότερο. Ε, ε, Πάνω απ' όλα, να πω ότι αυτό το κείμενο δρομολογείται πολύ γρήγορα. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το ρυθμό βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας. Μας συμφέρει όλους σαν κοινοβουλίο να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Να εγκριθούν οι νέες προδιαγραφές για την ασφάλεια των δικών μεταφορών. Βλέπουμε και από τα στατιστικά στοιχεία ότι απαιτείται κάτι τέτοιο που μας παρουσιάζει το Eurostat. Γενικά, επίτευξη των στόχων οδική ασφάλεια έχει υποστεί κάποια βιβράδυνση τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το πούμε. Για διάφορου λόγου. Άρα κατεπηγόντως απαιτείται αναθεώρηση τη οδηγία. Η αναθεώρηση είναι ευέλτιστο βήμα πρόοδου. Εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των οδικών υποδομών στην Ένωση και μέσω καλύτερης διαχείριση των διαδικασιών που ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Η πρόταση λοιπόν η αρχική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεωρώ ότι είναι καλή αφετηρία. Κυρίως όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Να συμπεριληφθούν οι αυτοκινητόδρομοι και οι πιο βασικοί δρόμοι που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Καλή και η προσέγγιση ενεργού, ενεργών λύσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες αξιολογήσεις ε, με βάση τα δεδομένα αντιδρώντας την κατάσταση. Όσον αφορά την ασφάλεια της υποδομής και καθέτος και οριζοντίως η σήμανση, προστασία των ευαλώτων χρηστών, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν και ενισχυθούν. Χρειάζεται καλύτερη ποιότητα σηματοδότησης και πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα γι' αυτό. Και τα ελάχιστα προαπαιτούμενα να καθοριστούν για τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα όσον αφορά και τις συσκευές που είναι πάνω στα αυτόματα οχήματα και που αφορούν τη χρήση των εφιών αυτοκινητοδρόμων. Λοιπόν, όσον αφορά το κείμενο που προτάθηκε, θα προτείνω και άλλες τροπολογίες ε, για, κάπου, για διεύρυνση της κάλυψης του τομέα. Άλλο θέμα που αφορά το πεδίο εφαρμογής. Ο τίτλος της ίσως να ξεγελά διότι εξετάζει τα θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια επιφανειακά. Ενώ στον τίτλο αφήνει να εννοηθεί κάτι άλλο. Συνδέεται με τα θέματα που αφορούν τι προδιαγραφέ διαδικασίε ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν προ βελτίωση τη κυκλοφορία ε, των οχημάτων και των οδηγών. Όμω το θέμα σταθερότητα των υποδομών θα έπρεπε να εξεταστεί, διότι αυτό επηρεάζει σημαντικά τον τομέα, όπως δυστυχώς είδαμε πρόσφατα με αυτά που συνέβησαν, τα σοβαρότατα γεγονότα που συνέβησαν στην Ιταλία. Γι' αυτό το λόγο, γνωρίζοντας ότι το θέμα δεν εξετάστηκε πραγματικά, θα ήθελα εντό προτάσεως να εισαγάγω κάποια στοιχεία. Και έτσι να εξετάζονται και οι υποδομές, να ελέγχονται όσον αφορά τις γέφυρες και τις σύραγγες χρησιμοποιώντας ε, καινοτόμε τεχνολογίες και μεθοδολογίες. Άλλο στοιχείο που έχει προτεραιότητα. Η προστασία των ευαλώτων χρηστών αυτοκινητοδρόμων. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Να βελτιώσουμε τους ελέγχους τη οδική ασφάλειας. Και να αξιολογηθούν οι δρόμοι στο επίπεδο των δικτύων. Πιο ενεργή συμμετοχή όλων των χρηστών. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη δική ασφάλεια να δημιουργηθεί ένα σύστημα σήμανσης εθελοντικής για να διευκολύνονται οι αναφορές ε, λεπτομεριών στον αφορά τους κινδύνους που υπάρχουν και τι θεωρούν ε, οι χρήστες των οχημάτων, οι οδηγοί, ε, ότι είναι σημαντικά θέματα ασφαλείας να αποφύγουμε ατυχήματα και να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία όταν αξιολογούμε την ασφάλεια. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια για τους χρήστες των οδών μέσω ενδείξεων στους δρόμους και των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Συνοπτικά αυτό είναι το προτινόμενο κείμενο. Είμαι στη διάθεση ε, των συναδέλφων που θα ήθελαν να κάνουν κάποιες προτάσεις και έχουν κάποιες εισηγήσεις να κάνουν. Ευχαριστώ κυρία Γιούτο. Ο κύριος Ντελή. Θέλετε να μιλήσετε? Είσαστε το αρχαιότερο μέλος ε, του ΕΛΚΑ και το πιο υψηλό βαθμό τροποντινά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η βοηθός κυρία Σμιτ μου ζήτησε να λάβω μέρος στη συζήτηση, γιατί η ίδια δεν μπορούσε να παραστεί, στον αρχηγέρος, και γι' αυτό θα διαβάσω τι μου έδωσε αισθάνομαι σαν παρουσιαστή ειδήσεων. Συγγνώμη γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το σκοπό αυτού του φακέλου, όλοι συμφωνούμε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να μειώσουμε του θανάτου στους δρόμους. Η ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί ε, τις τελευταίες δεκαετίες ε, και χάρη στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2001 μέχρι το 2010 ο αριθμός των θανάτων στους δρόμους ε, έπεσε κατά 43% και 19% επιπλέον από το 2010 μέχρι το 2016. Όμως το 2016 μόνο 25.620 άνθρωποι έχασαν το, τη ζωή τους από τροχέα. Ε, επίσης η επικουρικότητα και η ευθύνη. Ε, αυτό είναι κοινό στόχο. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι κατά ανάγκη ντε και καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να, κάνει, να αναλάβει θέσεις δράσεις. Ούτω ή άλλω οι άνθρωποι κάνουν και θα κάνουν λάθη. Είναι υπεύθυνοι όλοι οι φορεί σε όλα τα επίπεδα, ούτω ώστε τα ατυχήματα στον δρόμο να μην οδηγούν σε θανάτους. Ε, όσο, ακόμα και αν είναι υπερβολικά καλέ οι κατευθυντήριε γραμμέ μα. Όσο ωραία και αν διατυπώνουν οι γραφειοκράτες ε, τις διατάξεις αυτές της Βρυξέλλης, πάντα κάποιοι θα μεθάνε, θα είναι κουρασμένοι ενώ οδηγούν ε, και κάποιοι άλλοι κοιτάνε το κινητό τους ενώ οδηγούν. Επομένως, δεν έχει σημασία ποιος διατυπώνει τους κανόνες, εάν τα άτομα δεν τους ακολουθούν. Ω ΕΛΚ δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είναι αλήθεια βεβαίως ότι μόνο 8% των ε, θανατηφόρων τροχαίων έγιναν στα δίκτυα TNT. Όχι χάρη στην ε, καλή οδηγία, αλλά γιατί στις, ε, στους αυτοκινητοδρόμους δεν έχουμε ποδηλάτες, δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε πεζούς κτλ. Οι αυτοκινητόδρομοι είναι οδοί ταχείας κυκλοφορία για τη μεταφορά μας. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τα θαντιφόρα τροχέα, να, θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ε, περισσότερο του κινητοδρόμους παρά τους, ε, το δευτερεύον οδικό δίκτυο, δίκτυο το οποίο, ε, στο οποίο έχουμε περισσότερα ατυχήματα και μάλιστα μοιραία. Ε, τρίτον, οι νέε τεχνολογίες. Είμαι κατά της επέκτασης του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας, αλλά και γενικά το ΕΛΚ θέλει παρόλα αυτά να, συνεργασ... να συνεργαστούμε ε, για τη σήμανση στις, με τις πινακίδες, αλλά και τη σήμανση πάνω στο δόστρωμα ε, για τα φορτηγά κτλ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, και ότι έχουμε κατάλληλα ε, πρότυπα τα... αν έχουμε ενιαία πρότυπα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μόνο τότε πρέπει να βάλουμε αυτόνομα ε, κινούμενα οχήματα. Η η ευθύνη ε, για την ασφαλή κυκλοφορία ενός τέτοιου οχήματος δεν μπορεί να περάσει στους διαχειριστές ε, της ε, κυκλοφορίας. Ευχαριστώ κύριε Ντελή. Από τους σοσιαλιστές δεν υπάρχει άνθρωπος. Ο κύριος Ευχαριστώ συνάδελφοι. ευχαριστώ συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κυρία Ντανιέλα Αιούτο για την έκθεση αυτή. Θα μιλήσω γενικόλογα, θα κάνω γενικά σχόλια, γιατί το βασικό είναι ότι το περιεχόμενο της έκθεσης είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να είναι. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας και κυρίως για την ομάδα μου. Και είμαστε ικανοποιημένοι που ο αριθμός των μοιραίων τροχαίων ε, στους δρόμους μας τις τελευταίες δεκαετίες μειώνεται σταθερά. Παρ' όλα αυτά ε, έχουμε φτάσει ε, σε ένα επίπεδο και δεν μπορούμε να κατέβουμε τα τελευταία χρόνια από αυτό, να μειώσουμε ακόμα περισσότερο του θανάτου. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε πώ θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να προσαρμόσουμε την υποδομή μας στις εξελίξεις, σε όλα έχουν συμβεί πρόσφατα και να λάβουμε υπόψη μας τις νέες τεχνολογίες που μπαίνουν στη ζωή μας, νέα είδη οχημάτων και τη φύση των οδηγών που αλλάζει. Θα πρέπει να βελτιώσουμε ε, την συντήρηση των δρόμων επίσης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε σε πρακτικό επίπεδο τους δρόμους μας όπως μπορούμε και όσο μπορούμε. Δεν νομίζω ότι επίσης δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τους, τις ευάλωτες ομάδες χρηστών των δρόμων. Επίσης, ε, το φάσμα της, ε, των υπερβολικών κανόνων είναι τελείως λάθος ε, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές και άλλες και γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των διαφορών χωρών και διαφορετικές προποθέσει. Παραδείγματο χάρη διαφορετικές πινακίδες και σήματα στον, στο οδόστρωμα ε, αφορούν ε, συγκεκριμένους κινδύνους, συγκεκριμένες καταστάσεις ανάλογα με το που είσαι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια πράγματα παντού. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το δίκτυο TEN-T το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών δηλαδή και τις μεγάλες αρτηρίες ε, καθώς και τους δρόμους που συνδέουν ε, περιοχές πριν, να εστιάσουμε εκεί πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Θα στείλω τροπολογίες για να βελτιώσουμε αντιπεραιτέρω το κείμενο. Οποιοδήποτε θύμα στο δόστρωμα είναι μια τεράστια απώλεια θα πρέπει να κάνουμε το καταδύναμη, ούτω ώστε να μειώσουμε τα μοιραία τροχέα, τα θαντιφόρα τροχέα σε, στο μηδέν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μασμάκερ. Συνάδελφο και το λόγο. Από του σοσιαλιστέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρου του Ματέα. Δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα. Μου είπε να διαβάσω τη δήλωσή του. Ευπρόσδεκτη πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζω την, ε, αυτή την οδηγία και τους στόχους αυτής της πρότασης που στοχεύει στην μείωση των θρατηφόρων ατυχημάτων και των τραυματισμών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους ευάλωτου ε, χρήστε ε, τη οδική υποδομή. Και προφανώς η βελτίωση των υποδομών είναι σημαντική για τη βελτίωση τη ασφάλεια αλλά και την καλύτερη σύνδεση των, των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Υποστηρίζω την πρόταση τη Επιτροπής για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία πέραν των διευρωπαϊκών δικτύων. Κάτι τέτοιο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ε, ε, θα μπορούσε να υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα και γι' αυτό ε, θα θέλαμε ε, σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ε, να γίνει μια αξιολόγηση ε, αντικτύπου ακριβώ έτσι όπω προτείνεται και από, τον εισηγητή, επίσης, από την εισηγήτρια. Επίση, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί περισσότερο άχθο για τα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν αλληλεπικαλύψει, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι αξιολογήσει, σε ό,τι αφορά το σύνολο του οδικού δικτύου και τι δοκιμέ ασφαλεία. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζω την πρωτοβουλία για την αυξημένη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αναμένω με ενδιαφέρον τη μελλοντική μα συνεργασία και σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Δεν έχουμε άλλους εκπροσώπους των ομάδων. Θάρρο. Α, συγγνώμη. Ορίστε. Να θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ε, διάβασα πολύ προσεκτικά την πρόταση, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ε, υποδομή αφενός ε, και την εκπαίδευση των οδηγών αφετέρου. Γιατί από τις ε, μελέτες προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, τα ασφάλματα τα οποία διαπράττουν οι οδηγοί παίζουν συνεχίζουν να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από ότι η οδική υποδομή. Οπότε θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο έχει ληφθεί υπόψη αυτή η παράμετρο σε αυτή τη συζήτηση. Εκτό κι αν αυτό που αναφέρω τώρα, δηλαδή εκπαίδευση των οδηγών, δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη. Ευχαριστώ. Έχει θέση στη συζήτηση αυτό το θέμα. Η έκθεση επικεντρώνεται επί των υποδομών. Αλλά υπάρχει και διασύνδεση μεταξύ των υποδομών και της δυνατότητας διάπραξης φαλμάτων αλληλένδετα τα θέματα. Μιλάμε για ασφάλεια. Μετά τις υποδομές θα αναφερθούμε και στο πρόβλημα της οδήγησης. Θα δώσω το λόγο στην συγγήτρια μετά, στην ολοκλήρωση της συζητήσεως. Η κυρία Γιούτο μπορεί να πει κάτι πάνω σε αυτό. Να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την κυρία Ιωαννίδου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμε βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την συνεχή υποστήριξη του βασικού μας στόχου, δηλαδή τη ε, δραστική μείωση ε, του αριθμού των ατυχημάτων με θανάτους και ε, τραυματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντοτε ποιο είναι ο βασικό στόχο μα, αλλά ε, στη σήμερα ημέρα 25.000 άτομα ε, συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή του ετησίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 17 άτομα καθημερινά. Δηλαδή, σαν να μιλάμε ένα ολόκληρο λεωφορείο από ανθρώπου. Οπότε μιλάμε για ανθρώπου του οποίου θα λείψουν από τι οικογένειέ του και κατά συνέπεια θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα σε αυτό το φάκελο. Εδώ λοιπόν ο στόχος μας είναι μηδενική, ε, μηδενική θάνατο, μηδενικός αριθμός ε, θανάτων στο δικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050. Ε, και εδώ ε, η προσέγγιση μας εστιάζει φυσικά στα οχήματα και φυσικά και στους οδηγούς, αλλά και στην υποδομή που αποτελεί δηλαδή το τρίτο πυλώνα αν θέλετε Άρα λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του τρίτου πακέτου κινητικότητας το οποίο παρουσιάστηκε το Μάιο του 2018 η Επιτροπή ε, παρουσίασε ακριβώς μια τέτοια ολιστική σφαιρική προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου μας λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιμέρους ε, παραμέτρου. Η υποδομή λοιπόν είναι το αντικείμενο αυτής εδώ της πρόταση, γιατί στο 30% των θανατηφόρων ατυχημάτων ε, η υποδομή παίζει ένα ρόλο. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε την πρόταση για τροποποίηση της εφιστάμενης οδηγίας με τέσσερα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά αλλάζουμε σε αυτή την πρόταση. Το πρώτο είναι η βελτίωση της διαφάνειας αλλά και της, του follow-up, δηλαδή Τη συνέχεια που δίνουμε στι ε, διαδικασίε διαχείριση των κινδύνων. Ε, πρόκειται για μια οδηγία η οποία έχει λειτουργήσει καλά στο παρελθόν, αλλά ε, δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε ω προ το τι συμβαίνει ω συνέχεια των διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα. Από εκεί και μετά θέλουμε να προσθέσουμε μια ενεργό διαδικασία με βάση την οποία θα χαρτογραφούμε, αν θέλετε, την ασφάλεια σε όλο το οδικό δίκτυο. Και εδώ ακριβώ λέμε ότι είμαστε, δραστηριοποιούμαστε με δική μα πρωτοβουλία. Θέλουμε δηλαδή δηλαδή η αξιολόγηση να γίνεται εκ των προτέρων. Εκ Τρίτο στοιχείο είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία ε, πέραν των διευρωπαϊκών δικτύων σε όλε τι κύριε οδικέ αρτηρίε. Και το τέταρτο στοιχείο είναι η βελτίωση της, ε, των σχετικών επιδακίδων και τη σηματοδότηση. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στα ε, δύο στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν και στη συζήτηση εδώ. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την υποστήριξη που δείχνεται απέναντι στις ε, οδηγές πινακίδες και τα σήματα γιατί πραγματικά θεωρούμε πως θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην αυτοματοποιημένη αλλά και στην αυτόματη οδήγηση. Ήδη τη σήμερα ημέρα υπάρχουν διαφορετικά ε, επίπεδα αυτονομία του οχήματο και συστήματα που υποβοηθούν τον οδηγό. Για παράδειγμα, το σύστημα τη της παραμονή στην ίδια λωρίδα κυκλοφορία ή ε, το σύστημα ανάγνωσης ε, των ε, σημάτων κυκλοφορίας που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν την αποφυγή, στην αποφυγή ατυχημάτων. Άρα λοιπόν θεωρούμε πως με την περαιτέρω βελτίωση μπορούμε να επιτύχουμε ένα περαιτέρω όφελο αφού θα υπάρξει και περαιτέρω χρήση αυτών των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Ένα ακόμα, ένα ακόμα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε επανειλημμένα εδώ είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία πέραν των διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, να σα πω ότι ο στόχο μα εδώ πραγματικά είναι να εστιάσουμε στι κύριε οδικέ αρτηρίε, στου κύριου αυτοκινητοδρόμου. Δεν θέλουμε δηλαδή να επηρεάσουμε άλλε υπαρχιακέ όντω ε, δευτερεύουσα σημασία. Αλλά θέλουμε να καλύψουμε όλε εκείνες τις οδικέ αρτηρίες ε, όπως εκείνες που καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Και ο στόχο μα εδώ σήμερα ε, ε, και το βασικό μας σκεπτικό είναι ότι το δίκτυο ε, των ευρωπαϊκών δικτύων είναι το ασφαλέστερο γιατί στοιχεί στο 4% του, του συνολικού δικτύου και ευθύνεται για το 8% των θανάτων. Άρα λοιπόν αποφασίσαμε, να αποφασίσουμε να διαβρύνουμε αυτό το σύστημα θα μπορούσαμε να καλύψουμε το 15% του δικτύου αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε το 40% ε, των θανατηφόρων ατυχημάτων. Δηλαδή, μια σχετικά, σχετικά περιορισμένη αύξηση του πεδίου εφαρμογή πέραν δηλαδή των διευρωπαϊκών δικτύων και σε άλλε κεντρικέ αρτηρίε θα οδηγούσε σε σημαντική κάλυψη και μείωση δηλαδή των θανατηφόρων ατυχημάτων. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την έκθεσή τη, η οποία έχει ω στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των στοιχείων που προτείνει η Επιτροπή μέσω για παράδειγμα της ενίσχυσης ε, των δράσεων σε ό,τι αφορά ε, τα ευρωπαϊκά οδικά σήματα ε, και τις πινακίδες και μια αξιολόγηση ως προς τη σκοπιμότητα της ενδεχόμενης εναρμόνισης αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η πρότασή σας περιλαμβάνει περαιτέρω στοιχείο σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης όπως και η δυνατότητα για τους οδηγούς να κοινοποιούν ε, κινδύνου του οποίου οι ίδιοι εντοπίζουν ε, στον δρόμο. Θεωρούμε πω είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι προτάσει και θα θέλαμε να τι συζητήσουμε περαιτέρω. Ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την ε, προσοχή σα από την πλευρά τη Επιτροπή και το οποίο ανέφερε η κυρία Αγιούτο, δηλαδή υποχρέωση των κρατών μελών, ή υποχρεώσει του σε ό,τι αφορά την δομική αποτελεσματικότητα των ε, γεφυρών τους και των τούνελ τους σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα συντήρησης. Ναι, εδώ θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά ε, με βάση αυτή την προτινόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου τι εθνικέ αρμοδιότητε που ισχύουν σε αυτό το τομέα. Ε, Πάντω, σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να συζητήσουμε περαιτέρω του τρόπου για την επίτευξη και αυτών των στόχων και σα ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική μα συνεργασία. Ευχαριστώ, κυρία Ιωνίδου. Ο λόγος στην κυρία Γιούτο για να ολοκληρώσει το θέμα, την συγκεκριά μας. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτές τις σκέψεις. Ο συνάδελφος Βαντενκάπ βαίνω ότι απεχώρησε. Ήθελα να του πω μερικά πράγματα σχετικά με τις παρατηρήσεις του. Ο ανθρώπινος παράγων σαφώς είναι βασικός παράγων που οδηγεί στο ατύχημα πέρα από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι. Όμως η διεύρυνση καλύπτοντας όλα αυτά που αφορούν τις υποδομές, εγγυάται την ασφάλεια, που σημαίνει ότι μειώνεται το βάρος για τον οδηγό όταν οδηγεί. Άρα, εξ αυτού μειώνει και το ποσοστό ανθρωπίνου σφάλματος. Αυτό αναμένουμε από την εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια των υποδομών. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα να παρεύουμε επί της σταθερότητας και της ποιότητας των υποδομών. Δεν ήταν στο αρχικό όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργαζόμαστε όμως και αυτή κατά την άποψή μου είναι μια καλή ευκαιρία για να εισάγουμε κάποιο στοιχείο που θα φανεί χρήσιμο. Αν βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε και να μπορέσουν να παρέμβουν τα κράτη-μέλη χωρίς υπερβολικό βάρος και να αναλάβουν τις κατάλληλες ευθύνες θα είναι καλό για να αποφύγουμε τις καταστροφές που γνωρίζουμε. Λοιπόν, περιμένω τις τροπολογίες μας. 24 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία. Έχουμε σύντομο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 25 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. 25 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ήδη έχουμε προχωρήσει γρήγορα. Θα, τελειώσουμε σύντομα. Δηλαδή όσο προχωρούμε φεύγει και ο κόσμος. Η Κριστίν είναι στην αφετηρία. Τώρα, πρόταση κανονισμού σχετικά με το, το Ταμείο Συνοχής Η κυρία Μπονφουά λοιπόν έχει το λόγο που είναι η Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την έκθεση. Έχουν κατατεθεί καμία κατοστή τροπολογίες για αυτό το κανονισμό που πλαισιώνει την, ε, τον επόμενο προγραμματισμό του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξη. Οι τροπολογίε πήγαν προ την ίδια κατεύθυνση για να ενισχύσουν την ε, κατεύθυνση των μεταφορών και τις προτεραιότητε που είχαμε το, το, Τηθούν από αυτά τα Είμαι πεπισμένη μετά από την πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών που πήγε πάρα πολύ καλά την περασμένη εβδομάδα. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε καλέ συμβαστικέ τροπολογίε ε, μέσα σε αυτή την ε, πολύ σφιχτή προθεσμία που έχουμε. Σε ό,τι αφορά την ε, θεματική συγκέντρωση, έλαβα υπόψη τι διάφορε προσεγγίσει που προτείνουν οι βουλευτέ. Κάποιοι βουλευτές ε, θέλουν νέους στόχους ε, στη θεματική συγκέντρωση, ενώ άλλοι βουλευτές θέλουν να κατεβάσουμε το επίπεδο συγκέντρωσης ή να μην αγγίξουμε το κείμενο που προτείνει η Κομισιόν. Αφού ανάλυσα τις διάφορες απόψεις και άκουσα τις παρατηρήσεις κατά την παρουσίαση της εκθεσή μου, αντί να προσθέσουμε νέους στόχου, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση, κατεβάζοντας το επίπεδο συγκέντρωσης των πόρων προς τον πολιτικό στόχο υπαριθμών 1, δηλαδή μια Ευρώπη πιο έξυπνη, η οποία, κάτι που αφορά και το ψηφιακό πεδίο, για να δώσουμε περισσότερες ε, αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές για να χρηματοδοτήσουν και άλλους πολιτικούς στόχους, όπως τον στόχο 3, δηλαδή μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη ή τον ε, στόχο 4, μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, οδήγησε σε συμπεράσματα. Ε, θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Έχουμε μια δεύτερη συνεδρίαση σχεδόν εισηγητών ε, στην Ολομέλεια του Στρασβούρου και νομίζω θα φτάσουμε σε καλές προτάσεις από πλευράς Επιτροπής Μεταφορών. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ αισιόδοξα λόγια. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Ντελή, ο κύριος Μπά, Μπά από το ΕΛΚΑ. Ουδής, πολύ ωραία. πάλι ο κύριος Ντελή. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, με τιμή θα εκπροσωπήσω την κυρία Κλάουντια Μοντέρο αυτή τη φορά. Θα διαβάσω το μήνυμά της. Είναι μέρα ανάγνωση για μένα. Ένα-δύο σημεία η πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική γιατί κάνει επενδύσει, αλλά με τι ε, περικοπέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το, τα έτη 2021 έω 2026 υπάρχει κίνδυνο να ε, βαθύνουμε τι διαιρέσει στην Ευρώπη. Η σύγκληση, σταδιακή σύγκληση των λιγότερων επιτυγμένων περιοχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν πόσο σημαντικά είναι τα Ταμεία Συνοχή και το Ταμείο Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη για να μειωθούν οι ανισότητε στην Ευρώπη. Τρίτον, για αυτού του λόγου η εισηγήτρια είναι υπέρ σκιώδη είναι υπέρ της δυνατότητα υποστήριξης των επενδύσεων στα αεροδρόμια, ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές. Ε, Έχουμε το άρθρο 349 για αυτές τις περιοχές ε, στη συνθήκη, όπου έχουμε 9 περιοχές βασικά, λόγω των ε, δομικών, κοινωνικών ε, συνθέσεών τους, θα πρέπει να έχουν ειδικά μέτρα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα διορθωτικά ταμεία. Οι περιοχές αυτές σας, επίσης, με βάση την τρέχουσα νομοθεσία, θα πρέπει να λάβουν υποστήριξη για επενδύσεις, για την αντιμετώπιση των υπολοιμάτων των αποβλήτων δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι 8 από τις 9 νησιωτικές περιοχές, από τις 9 περιοχές είναι νησιωτικές και θα πρέπει να συμπληρώσουμε το κόστος που θα αναλάβουν αυτές οι περιοχές. Η θεματική συγκέντρωση για αυτές τις περιοχές, άρθρο 3, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί. Οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικά στοιχεία συνοχής ε, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα αν η Ένωση πραγματικά υποστηρίξει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Τέταρτο σημείο για τις χώρες που υποφελούνται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, η θεματική συγκέντρωση και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτες. Και το μερίδιο για τη θεματική συγκέντρωση για τους πολιτικούς στόχους, στόχους πολιτικής παριθμών 1 και 2 θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερη από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Η ευελιξία για τις ε, περιφέρειες αυτές σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αυτούς τους στόχους ε, στις πολιτικές που θεωρούν καλύτερο αντί να έχουμε ελάχιστο μερίδιο για τη θεματική συγκέντρωση για όλους τους στόχους πολιτικής, αυτό σημαίνει, αν κάνετε αυτό που λέω, σημαίνει λιγότεροι, α, λιγότεροι κανόνες και εφαρμογή σε διάφορα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά το πεδίο υποστήριξη άρθρο 4 για το ERDF και το Ταμείο Συνοχής στο άρθρο 5, ε, θέλουμε ξεκάθαρα σημεία με τη δυνατότητα υποστήριξης υποδομών αεροδρομίων ε, και εξοπλισμών. Ε, κάναμε μία ε, συνάντηση των σχεδόν εισηγητών ήδη για τα γενικά θέματα και η επόμενη συνάντηση θα είναι στο Στρασβούργο, όπου θα ξανασυζητήσουμε. Αυτά είναι τα σημεία της κυρίας Μοντέρο. Ευχαριστώ κύριε Ντελή. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Η κυρία Μάισνερ από τους φιλελεύθερους όμως έχει το λόγο. Ναι, ξανά εγώ και εγώ θα διαβάσω μια δήλωση από τον συνάδελφο Τέλισκα, δηλαδή όπως και ο συνάδελφο Τέλη και εγώ διαβάζω μενούματα σήμερα. καταρχήν ευχαριστούμε λοιπόν για αυτό το σχέδιο και ε, ζητά συγγνώμη ο συνάδελφο που δεν βρίσκεται εδώ. Πάντω ε, είναι πολύ σύντομη η τοποθέτηση γιατί συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τα όσα προτείνει ε, ο εισηγητή και γι' αυτό δεν έχει υποβάλει και τροπολογίε. Υποστηρίζει δηλαδή την καλύτερη συμπερίληψη των στόχων που αφορούν δικότερα στις ε, μεταφορές ε, μέσα στους γενικότερους στόχους ε, και εξεπλάγει με το γεγονός ότι η Επιτροπή αναφέρει μόνο στο πίο 2 της μεταφορές και όχι στο πίο 3 σε ό,τι αφορά δηλαδή, την ενεργειακή μετάβαση. Οι βιώσιμη τρόποι μεταφορών είναι αποτελεί έκπληση ότι δεν συμπεριληφθήκαν ε, υπόψη υπό αυτή την προτεραιότητα. Επίση, ο κύριο ε, Τέλισκα προτείνει την ε, καλύτερη παρακολούθηση του προγράμματο και αναμένει με ενδιαφέρον τι συναντήσει των σχεδόν εισηγητών. Πάντω, υπάρχει ένα σημείο επί το οποίο διαφωνεί με τον εισηγητή, όπω το κοινοποίησε κατά την τελευταία συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Δηλαδή, η χρήση των ERDF και του Ταμείου Συνεχή σε ό,τι αφορά την αγορά του Rolling Stock για του σιδηροδρόμου. Δηλαδή, δεν υποστηρίζει αυτήν την πρόταση συμβιβασμού κύριο κύριος σε ό,τι αφορά δηλαδή τις αγορές ε, ε του τροχαίου υλικού. Ευχαριστώ κυρία Μεσνέρ. Από τους πράσινους, ντεποντή, κανένας. Η κυρία Γιούτο, δεν θέλει να μιλήσει. Όχι. Τρομακτικό είναι. Από τους αριστερούς στην ΚΟΕ, ουδής. Από την Κομισιόν υπάρχει εκπρόσωπος. Υπάρχει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και έχετε το λόγο. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Για το σχέδιο γνωμοδότησης, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την δουλειά που έκανε βεβαίως. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που προτείνει η Κομισιόν στο άρθρο 2 για τους ειδικού στόχους και στο άρθρο 4 για το πεδίο εφαρμογή. Η πρόθεσή μας ήταν να διδαχτούμε από την περίοδο 2014-2020 και να κρατήσουμε την περιγραφή των στόχων και το πεδίο εφαρμογή σύντομα, σύντομ, σύντομες και απλές και για να εξασφαλίσουμε επαρκή ευελιξία σε επίπεδο προγραμματισμού αλλά και εν μέρη για να αποφύγουμε αυτό που συνέβη σε κάποιο βαθμό στην προηγούμενη περίοδο, δηλαδή 14-20, όπου καταλήξαμε με υπερβολικά μακροσκελή περιγραφή και κατάλογο α, πιθανού περιεχομένου παρά, ε, σύντομων, παρά σύντομους στόχους. Εξού και η περιγραφή που έχουμε λοιπόν. Τώρα, τι προσπαθήσαμε να πετύχουμε με τη θεματική συγκέντρωση. Έγιναν πολλές συζητήσει για το αν η θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο ή όπως γίνεται σήμερα σε περιφερειακό επίπεδο. Η άποψη της Κομισιόν ήταν ότι με το να έχουμε θεματική συγκέντρωση και ποσοστά θεματική συγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο προσφέρεται μεγαλύτερη ευελιξία σε περιφερειακό επίπεδο τελικά. Γιατί δεν χρειάζεται κάθε περιφέρεια ας πούμε, να ε, σεβαστεί το ίδιο ποσοστό όπως γίνεται σήμερα ε, γιατί έχουμε αυτό το στοιχείο σε περιφερειακό επίπεδο για το, την περίοδο 14-20. Επομένως, ε, έτσι επιτρέπουμε διακυμάνσεις από περιοχή σε περιοχή, περιφέρεια σε περιφέρεια ανάλογα με τις ανάγκες ε, της εκάστοτε περιφέρειας. το δεύτερο στοιχείο για τη θεματική συγκέντρωση είναι ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνε της Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάζουν στις βασικές ενωσιακές προτεραιότητες. Αυτές οι προτεραιότητες είναι το κλίμα και η καινοτομία. Υπάρχει επαρκής ευελιξία στην πρόταση και για άλλους τομείς μπορούμε να το στοχεύσουμε και οι περιφέρειες και τα κρατημέλη μπορούν να ξοδέψουν και σε άλλου τομεί, αλλά για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη από τι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ποσά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να επικεντρωθούμε στη συγκέντρωση στο κλίμα και την καινοτομία. Και για λόγου συνέπειε επίση, αλλά και για να ευθυγραμμιστούμε με τι ενωσιακέ προτεραιότητε, προσπαθούμε, ειδικά στο άρθρο 6, να ευθυγραμμίσουμε να θυραμιστούμε με τις αρνητικές προτεραιότητες, δηλαδή η διατύπωση για τον αποκλεισμό που περιλαμβάνει, τις αποκλήσεις μάλλον που έχει το άρθρο 6, ε, ε, είναι θυγραμμισμένο με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές, για τα απόβλητα, ας πούμε, για την ε, ευρεία ζώνη και την ευρυζωνικότητα. προσπαθήσαμε να διδαχτούμε από την εμπειρία μας μέχρι τούδε, εξού και ο αποκλεισμό των υποδομών των αεροδρομίων που βασίζεται ας πούμε στις αρνητικές εμπειρίες που είχαμε στο παρελθόν ειδικά από την έκθεση ας πούμε, που ετοίμασε το ελεγκτικό συνέδριο πριν από 2-3 χρόνια και που μίλησε για αυτό το θέμα των αεροδρομίων. Ε, αυτό, είναι, αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο μετά το 2020. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Η συγγήτρια όχι εσεί πρώτα, ξέρω ότι έτσι δεν ήθιστε. Μετά την Κομισιόν κανονικά εσεί μιλάτε, αλλά πρώτα η κυρία, η συνάδελφό σα θα μιλήσει, η κυρία Ντεμόντι. Μετά. Θέλω να σα πω ότι γενικά συμφωνώ. Συμφωνώ σε εν πολλής με την πρόταση τη εισηγήτρια και εγώ θέλω να τονίσω τη σημασία του να κινηθούμε προ μια περιφερειακή κατεύθυνση παρά εθνική. Θέλουμε να δώσουμε βεβαίω προτεραιότητε. γιατί έχουμε μια πολύ διαφοροποιημένη η ευρωπαϊκή πραγματικότητα από κράτο σε κράτο. Ακόμα και στο εσωτερικό μια χώρα ε, υπάρχουν διαφορέ από περιφέρεια σε περιφέρεια. Νομίζω ότι τα ταμεία λοιπόν και τα κονδύλια του θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτό το στοιχείο, τη διαφορά αυτή που υπάρχει και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Λοιπόν, τώρα για τι μεταφορέ. Δεν συμφωνώ με τη γραμμή του να τιμωρήσουμε ας πούμε, τα περιφερειακά αεροδρόμια. Γιατί πρέπει να είμαστε πιο κοντά στην ε, πραγματικότητα ε, των εδαφών μας και σε αυτούς που δεν ε, είναι καλά συνδεδεμένοι. Και επίσης, αν βοηθήσουμε τα περιφερειακά αεροδρόμια, θα αποσυμφορήσουμε τα κεντρικά δεν λαμβάνεται υπόψη μα ότι υπάρχει διαφοροποιημένη πραγματικότητα, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο πολύ παρόντε στι στις διάφορες περιοχές, όχι μόνο στα μεγαλαστικά κέντρα και θα πρέπει να μειώσουμε τη συμφόρηση των μεγάλων αεροδρομίων κτλ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα έλεγα να υποστήριξουμε περισσότερο τα περιφερειακά αεροδρόμια, αντίθετα από αυτό που λέει η Κομισιόν, ε, και τι πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Μην, να μην λάβουμε υπόψη μας μόνο τις α, εξόχως απόμακρε περιοχές, αλλά και τις υπόλοιπες. Θα πρέπει να τους δώσουμε υπηρεσίες ούτως ώστε να αναπτυχθούν, πέρα από τον τουρισμό. Το είδαμε τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη μα τα όσα είπε το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά τι τρευλώσει. Πρέπει να αποφύγουμε βεβαίω. Αλλά το να φτάσουμε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές θα δώσουμε τη δυνατότητα στις πιο φτωχές περιφέρειες που χρειάζονται ανάπτυξη να αναπτυχθούν. Να υπάρξει εκεί μια οικονομία η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί. Ε, ο τριτογενής κλάδος οικονομίας δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Η συγκήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι σκιώδεις ηγητές των ομάδων και εγώ ανταλλάξαμε απόψεις επικοδομητικά. Και νομίζω ότι αυτό που αναφέρθηκε από τους ομιλήσαντες για το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι πρέπει να τονίσουμε ότι οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δράσουν άμεσα βάσει των προτάσεων που γίνονται και όχι μόνο μέσω με, μηχανισμού ευελιξίας σε επίπεδο κατών μελών. Δεν είναι η πρώτη έκθεση που βλέπουμε ότι συνεργάζονται οι ευρωβουλευτές με την τοπική αυτοδιοίκηση και επεξεργαζόμαστε και τις προτάσεις σχετικές επιτροπής των περιφερειών. Και θα συνεχίσουμε να το εφαρμόζουμε αυτό. Άκουσα τα διάφορα επιχειρήματα που αφορούν τις υπερπεριφερειακές περιοχές. Δεν μπορώ παρά να είμαι ευαίσθητη σε αυτό. Πρέπει να τονίσουμε αυτή την πτυχή. Να ενθαρρύνουμε ό,τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τις μεταφορές σε αυτές τις απομακρυσμένες περιφέρειες. Όμως όσον αφορά το τροχαίο υλικό πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο, διότι πολύ συχνά οι περιφέρειες είναι εκείνες που πρέπει να αγοράσουν το τροχαίο υλικό για τις κοινέ μεταφορές και επειδή αυτό επισέρχεται στις καθοριστήσεις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου θα πρέπει να συνοδεύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό. Την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση των σκιωδών θα καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα. Είμαστε φιλόδοξοι σχετικά με το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις περιφέρειες που πρέπει να παρεμβαίνουν πρώτες σχετικά με τον τομέα των μεταφορών. Α, συγγνώμη. Κάτι ξέχασα Όσον αφορά τους αερολιμένες και τις σχετικές υποδομές, το ίδιο ισχύει. Σε πρώτη γραμμή είναι ε, οι περιφέρειες και δεν θέλουμε να εξαιρεθούν από τον όλο μηχανισμό και να τις στηρίζουμε για να εξασφαλίζουμε ότι τα αεροδρόμια να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, χρηματοδοτηθούν σε επίπεδο περιφερειών και κρατών και να μην έχουμε υποδομές ε, που προέρχονται από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα αεροδρόμια και πρέπει πάνω σε αυτό να είμαστε άγρυπνοι φρουροί. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου στην Επιτροπή και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν από αυτή την ημερομηνία. Αντίθετα, από τους σιδηροδρόμους, εμείς είμαστε πιο μπροστά όσον αφορά το ωράριό μας. Έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου. Ίσως μπορούμε να συνεχίσουμε την πρόοδό μας αυτήν. Και να ζητήσουμε τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου, αν έχει την καλοσύνη, να έρθει εδώ και να μας κάνει την παρουσίασή του σχετικά με τα τρένα υψηλής ταχύτητας και το σχετικό σιδεροδρομικό δίκαιο, δίκτυο. Συγγνώμη. Euh, Ευχαριστώ τον κύριο Έριξ που εκπροσωπεί το ελεκτικό συνέδριο. Συστατικό σχεδιασμό όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των γραμμών των τρένων υψηλή ταχύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα ενδιαφέρον και σημαντικό. Δεν έτυχε πάντα τη δέουσα προσοχή. Η πραγματικότητα στην Ευρώπη χρήζει μια τέτοια εξέταση. Έχετε το λόγο λοιπόν για τη διάρκεια που επιθυμείτε. Σε ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ανταποκριθούμε λοιπόν σε αυτή τη φήμη που έχουμε, το ότι είμαστε πολύ ακριβείς και επιμελείς Είμαστε λοιπόν νωρίτερα από την ώρα μας εδώ και θα ξεκινήσουμε την έκθεσή μας αυτή σε σχέση με το δίκτυο το σύνδρομικό υψηλής ταχύτητας, ε, ποια ήταν τα πορίσματά μας και βέβαια είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήματα γιατί ε, προβήκαμε σε αυτόν τον έλεγχο. Υπήρχαν σημαντικοί κίνδυνοι σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση σε σχέση με τα τρία E όπω τα λέμε στα αγγλικά, δηλαδή ε, την οικονομία, την αποτοπικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ε, δηλαδή εκείνο που διαπιστώσαμε ή θέλαμε να δούμε κατά πόσο είναι το κόστος υψηλό και πράγμα το διαπιστώσαμε σε σχέση με το αποτέλεσμα αυτών των ε, δικτύων υψηλή ταχύτητα. Ε, και επίση είδαμε ότι υπάρχουν μια σειρά από υπερβάσει των σχετικών δαπανών, καθυστερήσει, ενώ ε, η αποτελεσματικότητα είχε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου αλλά και σε ό,τι αφορά τη μείωση των συμφορήσεων στα σημαντικά δίκτυα. Ε, πέραν αυτού, εκείνο που μας απασχόλησε ήταν η χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο του 2000 έως 2020. 23,7 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αυτά τα δίκτυα ε, υψηλή ταχύτητα και συμπληρωματικά 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στην δημιουργία των συστημάτων διαχείρισης, των ευρωπαϊκών συστημάτων Διαχείρισης της συνδρομική κυκλοφορία και το μεγαλύτερο ε, κομμάτι αυτών των κοντιλίων προήλθε από την ε, κοινή διαχείριση, το 62%. Και αν δούμε δηλαδή και εδώ αυτή την πίτα πάνω δεξιά το διάγραμμα, θα ε, δούμε δηλαδή την κατανομή ένα κράτο μέλο. Η Ισπανία λοιπόν απορρόφησε σχεδόν το ίμιση αυτών των χρηματοδοτικών κοντιλίων. 47,3%. και μετά από την ολοκλήρωση όλων αυτών των επενδύσεων ο στόχος είναι η Ισπανία να διαθέτει το δεύτερο ε, μεγαλύτερο συνδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας ε, στον κόσμο μετά από την Κίνα. Ε, τι ε, συμπεριλάβαμε λοιπόν στην μελέτη μας εδώ. Εξετάσαμε 10 ε, γραμμές υψηλής ταχύτητας και συμπληρωματικά 4 διασυνοριακές συνδέσεις ενώ και 30 ε, σύγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα για την περίοδο του 2020 έως 2013. Με αυτόν τον έλεγχο λοιπόν καλύψαμε περισσότερα από 5.000 5.000 χιλιόμετρα γραμμών ή το 50% των γραμμών υψηλή ταχύτητα τα οποία είτε βρίσκονταν ήδη σε λειτουργία είτε βρίσκονταν υποκατασκευή. Εδώ λοιπόν στον χάρτη βλέπετε σε πράσινο χρώμα τα ε, κράτη-μέλη εκείνα τα οποία καλύψαμε με αυτούς τους ελέγχους μας, δηλαδή εκεί όπου κάναμε τις επισκέψεις μας, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και Πορτογαλία. Σε αυτά τα έξι χρόνια λοιπόν συγκεντρώνονται το 84% ε, των ε, κονδυλίων της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είχαν το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη απορρόφηση. Ε, τώρα, περνάω στα πορίσματά μας, στις διαπιστώσεις μας. Καταρχήν σε ό,τι αφορά ε, τον τομέα της ε, στρατηγικού σχεδιασμού και της ε, λήψης των αποφάσεων. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ρεαλιστικό μακροπρόθεσμο σχέδιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου υπάρχει δεν βασίζεται σε μια αξιόπιστη ανάλυση. Και γι' αυτό θεωρούμε πως ο τριπλασιασμός του μήκους των γραμμών σε πάνω από 30.000 χιλιόμετρα έως το 2030, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 9.000, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει σήμερα. Ούτε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε οι συντονιστές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν τα απαραίτητα νομικά εργαλεία, τις απαραίτητες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά το επίπεδο λήψης των αποφάσεων για τα διασυνοριακά έργα. Και έτσι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη ε, με τα οποία έχει γίνει συμφωνία σε ό,τι αφορά την κατασκευή των σχετικών γραμμών προβαίνουν σε αυτές τις κατασκευές και κατά συνέπεια ε, δεν δημιουργείται έτσι ένα δίκτυο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης απλώς όπως αναφέρεται και στον τίτλο της έκθεσής μας ένα αναποτελεσματικό μόρφωμα αν θέλετε από κατακαιρματισμένο όμω τελείω μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών δηλαδή γραμμές σε εθνικό και μόνο επίπεδο κατακαιρματισμένος πράγμα το οποίο οδηγεί σε κακές διεθνείς συνδέσει. και δεν επιτυγχάνει την απαραίτητη υπεραξία που θα έπρεπε να προκύπτει από τέτοιου είδου συγχρηματοδοτούμενε ευρωπαϊκέ επενδύσει. Και να σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε τι ακριβώ εννοούμε. Ε, σε ό,τι αφορά την σύνδεση καταρχήν Μόναχο-Βανώνα και την ε, τη σχετική σύρακα από την οποία περνάει η εν λόγω ε, ε, σύνδεση. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικές, διαφορετικά χρονοδιαγράμματα από τα διαφορετικά κράτη-μέλη και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν συμφορήσεις έως το 2040 σε αυτές τις συνδέσεις. Δηλαδή θα, θα διαρκέσει ένα τέταρτο του αιώνα μέχρι του να υπάρξει πραγματικά αποτελεσματική ε, μεγάλη υπεραξία από αυτά τα κονδύλια τα οποία εγκρίθηκαν συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, έφτασαν στο ύψο το 58. Δεύτερο τώρα παράδειγμα που θα ήθελα να δώσω είναι η σύνδεση υψηλής ε, ταχύτητας μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, ειδικότερα Μαδρίτης και Λισαβόνας. 436 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για αυτό το έργο και κατά την, ε, το έτος 2016 και 2017 η κατασκευή από την πορτογαλική πλευρά είχε ξεκινήσει ενώ η κατασκευή ε, στην ισπανική πλευρά είχε σταματήσει 6 χιλιόμετρα πριν από το να φτάσει στα σύνορα. Και όπω βλέπετε δηλαδή εδώ στην φωτογραφία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνδρομική σύνδεση υψηλή ταχύτητα ανάμεσα στην ε, Πορτογαλία και την Ισπανία. Αυτό λοιπόν μα οδηγεί σε αυτή τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει ε, ένας ενιαίος σχεδιασμός, υπάρχει απλά κατακαιρματισμό σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό μεταξύ των κρατών μελών. Ε, να αναφερθώ όμω στι σχετικέ συστάσει τι οποίε κάνουμε σε σχέση με αυτά τα προβλήματα Προτείνουμε λοιπόν στην Επιτροπή να αποφασίσει ένα σχέδιο εκτέλεσης το οποίο θα είναι ρεαλιστικό και θα είναι εκτελέσιμο, σε, ε, εκτελέσιμο μακροπρόθεσμα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναδιατυπώσει τον σχετικό κανονισμό τα διευρωπαϊκά δίκτυα έτσι ώστε να ε, παρακολουθεί και να επιβάλλει ε, την έγκαιρη κατασκευή των σχετικών γραμμών υψηλή ταχύτητα. Ε, και επίση θεωρούμε πω ο κανονισμό ΕΦΑ από την Επιτροπή αλλά και από τα κράτη-μέλη θα πρέπει από κοινού να συνοδευτεί από καλύτερα εργαλεία εφαρμογή στην πράξη έτσι ώστε να επιταχυνθεί η εκτέλεση των έργων για τα οποία έχουν δεσμευθεί τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και νομίζω πως ε, προς αυτή την κατεύθυνση ήδη έχει, κάνει, έχει αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία Επιτροπή. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στο δεύτερο κομμάτι, αν θέλετε, δεύτερη ενότητα απορρισμάτων σε ό,τι αφορά την προετοιμασία και την εκτέλεση. Δεν υπάρχει λοιπόν παρκή ποιότητα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών σε ό,τι αφορά συνδέσει υψηλή ταχύτητα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, οι αποφάσει λαμβάνονται στα κράτη-μέλη με βάση πολιτικές εκτιμήσεις, ε, πολιτικούς παράγοντες και όχι μία εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αξιοποιούνται με τον αποτελεσματικό τρόπο ε, τα κονδύλια και δυστυχώς αυτό είναι ο κανόνας και όχι εξαίρεση, δηλαδή αναποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων. Υπήρξαν από εκεί και μετά καθυστερήσεις ε, των ε, έργων ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεκαετής και αυτό αφορούσε το ίμιση των έργων αυτών για παράδειγμα από τα 15 είχαν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις ενώ σε ό,τι αφορά τις 10 αυτές γραμμές φτάσαμε σε ε, υπερβάσεις του κόστους της τάξης του 25, των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σε ύψος 78% σε, σχέση, σε σύγκριση με τον αρχικό προπολογισμό. Πράγμα βέβαια το οποίο ε, βασίζεται εδώ η υπέρβαση δηλαδή, του κόστου στον εθνικό προϋπολογισμό. Επίσης διαπιστώσαμε ε, ότι το κόστος για αυτές τις ε, γραμμές είναι υπερβολικά ε, υψηλό, υπερβολικά Δηλαδή μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο με βάση τις 10 σύνδεσεις που ελέγξαμε. Και διαπιστώσαμε ή υπολογίσαμε ποιο είναι το κόστος το οποίο εξοικονομούμε σε κάθε λεπτό ε, κατασκευής στι γραμμέ, το οποίο ανέρχεται σε 90 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στι θετικέ εκτιμήσεις. Επίσης, ε, διαπιστώσαμε ότι η μέση ταχύτητα των εν λόγω, στις εν γραμμές ανέρχεται σε 45% της ε, ε, μέγιστη ε, δυναμικότητα, δηλαδή τη μέγιστη ταχύτητα που θα μπορούσαν να αναπτύσσουν τα τρένα σε αυτήν την ε, γραμμή. Που σημαίνει ότι δεν είναι παντού απαραίτητο η τέτοιου είδους σύνδεση και αυτό θα οδηγούσε βέβαια και σε πολύ σημαντικές εξοικονομήσεις. και θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, να γίνει μια αναβάθμιση των υφιστάμενων σειροδρομικών γραμμών, έτσι ώστε δηλαδή να καλυφθούν σχετικές ανάγκες. Και για να πούμε και ένα θετικό παράδειγμα, ε, στην σύνδεση μεταξύ Βενετίας και στην ε, ε, υπήρξε μια αναβάθμιση, ανακατασκευή, δηλαδή μετασκευή του υφιστάμενου συνδρομικού δικτύου, το οποίο οδήγησε σε εξοικονόμηση των σχετικών δαπανών κατά 5,7 δισεκατομμύρια ε, ευρώ με μείωση ή μάλλον ε, με αύξηση του σχετικού χρόνου ταξιδιού κατά μόνο 10 λεπτά. Δηλαδή ε, τόσο σημαντική εξοικονόμηση 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ με απλά και μόνο αύξηση του χρόνου ταξιδιού κατά 10 λεπτά. Αυτό είναι λοιπόν ένα παράδειγμα το οποίο θα έπρεπε να αναγνωριστούν και άλλα κράτη-μέλη. Τι λέμε προ την Επιτροπή τώρα, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε προποθέσει σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των έργων, για παράδειγμα αξιολόγηση των αναγκών σε ό,τι αφορά την κατασκευή γραμμών υψηλή ταχύτητα. Θα πρέπει δηλαδή ειδικότερα ε, project ή ε, έργα που είναι ψηλής προτεραιότητας να αντιμετωπίζονται και ως τέτοια. Και επίσης ε, θα πρέπει να ελέγχεται και να παρακολουθείτε ως προϋπόθεση και επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων. Επίσης, θα πρέπει η κατασκευή σε διασυνοριακά έργα να γίνεται ε, με, πιο, με λιγότερο γραφειοκρατικό άκτος, ε, ειδικότερα δηλαδή διακασίες για την, πρόσκληση, για την υποβολή ε, προσφορών είναι υπερβολικά περίπλοκες και θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθούν και για τον ίδιο λόγο one-stop shop έτσι ώστε να γίνονται ευκολότερα οι σχετικές διατυπώσεις. Τώρα περνάω στην τρίτη ενότητα των συστάσεών μα ή των παρατηρήσεών μα σε ό,τι αφορά την οπτική γωνία του πολίτη, δηλαδή ποιε είναι οι υπηρεσίε τελικά που παρέχονται στου ε, πολίτε σε ό,τι αφορά ε, τη διάρκεια του ταξιδιού, σε ό,τι αφορά το κόστο του ταξιδιού, σε ό,τι αφορά τι δυνατότητε κράτηση των εισιτηρίων. Εδώ διαπιστώσαμε ότι προφανώ είναι υψηλότερη ταχύτητα οι υφιστάμενε ε, γραμμέ, αλλά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τι εναέρειε κυκλοφορίε. Γιατί όταν θέλει κανεί να μεταβεί, για παράδειγμα, από το Μιλάνο στη Βαρκελόνη, στο Μόναχο, δηλαδή σε μεγάλες ε, ε, υπάρχει δυναμικό να ανταγωνιστούν οι συνδρομικές γραμμές της ε, ε, μεταφορές ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με τον συνολικό χρόνο του να φτάσει δηλαδή κανείς από τη μία πόλη στην άλλη. Ωστόσο διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τα συστήματα κράτηση στο σιδηρόδρομο σε σύγκριση με τι ενέργειε κυκλοφορία. Και επίση δεν γίνεται κατάλληλη συλλογή των πληροφοριών σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τη χρονική, δηλαδή την τήρηση των ωραρίων και επίσης δεν, υπάρχει και, δεν υπάρχουν δεδομένα τυποποιημένα σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των πελατών. Και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αντίστοιχε συστάσει στην Επιτροπή. Δηλαδή θα πρέπει να παράσχει ε, υποστήριξη στα κράτη-μέλη ώστε να υπάρξει ε, ένα ε, ενιαίο σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων, single e-ticketing, στο οποίο προφανώς θα συμπεριλαμβάνονται και γραμμές υψηλής ταχύτητας. Επίσης και οι πληροφορίες προς τους ε, πολίτες θα πρέπει να βελτιωθούν, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ετήρηση των ωραρίων, σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των πελατών και ό,τι καθεξής. Και φτάνω στην ε, τελευταία ενότητα, στο τελευταίο τομέα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εξέταση εδώ της Αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει επαρκή σε βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των επενδύσεων στο δίκτυο υψηλή ε, ταχύτητα μετά από την κατασκευή αυτών των γραμμών. Δηλαδή διαπιστώσαμε ότι οι... υπάρχουν λιγότεροι ταξιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις γραμμές ε, και μάλιστα ε, αυτός ο αριθμός βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από το benchmark, δηλαδή από εκείνο τον στόχο που είχε θέσει η ε, ε, επιτροπή σε ό,τι αφορά δηλαδή τα 9 εκατομμύρια ε, ταξιδιωτών. Διαπιστώσαμε δηλαδή πως το 50% των γραμμών ο αριθμός των ταξιδιωτών είναι χαμηλότερος. Αυτό οδηγεί στον κίνδυνο του ότι να αξιοποιούνται αναποτελεσματικά τα κονδύλια που επενδύθηκαν και συγκεκριμένα σε αυτές τις τρεις γραμμές που είχαμε πολύ χαμηλά επίπεδα ταξιδιωτών. Δηλαδή μιλάμε για κονδύλια 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, επίσης διαπιστώσαμε ότι και στις ε, ε, γραμμές οι οποίες κατασκευάζονται τώρα δεν βλέπουν να υπάρχει ε, δυναμικό και προοπτικές σε ό,τι αφορά δηλαδή, την αύξηση των ταξιδιωτών, των επιβατών. Ε, και αυτό οφείλεται και στο γεγονό ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων γραμμών. Δηλαδή, ακόμα ε, υφίστανται 11.000 εθνικέ διατάξει, ε, παρότι υπήρξαν ήδη από το 2010 συστάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να παραμεριστούν όλες αυτές, όλα τα εθνικά προβλήματα λόγω των εθνικών διατάξεων. Επίση, δεν υπάρχουν κοινέ διατάξει σε ό,τι αφορά έναν κοινό ανταγωνισμό, ένα κοινό δίκτυο ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τι γραμμέ υψηλή ταχύτητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία ή ανάμεσα στην Ιταλία την Αυστρία θα πρέπει τα τρένα να σταματάνε και να γίνεται μετεπιβίβαση με ε, ε, αποτέλεσμα βέβαια ο χρόνο με τον οποίο κερδίζουμε μέσω ακριβώ των τρένων υψηλή ταχύτητα να χάνεται λόγω αυτών των μετεπιβάσεων. Ε, Επίση, ο τρόπο αξιοποίηση αυτών των γραμμών είναι πολύ ε, περίπλοκο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη σχετική αγορά σε όλα τα κράτη-μέλη. Το διαπιστώσαμε ιδιαίτερα αυτό στην Γαλλία και την Ισπανία. Και επίση υπάρχουν άνηση όρια ανταγωνισμού σε σύγκριση ε, με άλλου μεταφορικού ε, φορεί, ε, για παράδειγμα ε, τις οδικές μεταφορές. Δηλαδή και η αρχή των, ε, του, του, ο υπεύθυνο πληρώνει, αλλά και σε ό,τι αφορά την επιβολή τελών δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η απαραίτητη ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για να πετύχουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα. Ε, περνάμε στι τρει τελευταίε λοιπόν συστάσει, τι οποίε δώσαμε στην Επιτροπή. Θα πρέπει να εξαλείψει λοιπόν η Επιτροπή όλα τα ε, διοικητικά και ε, ρυθμιστικά εμπόδια σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα των γραμμών. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν τα υπάρχει εκτέλεση από την βράδυ των κρατών μελών των διατάξεων προκειμένου ε, η, τα σχετικά τέλη σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο να είναι ισορροπημένα και επίσης ε, καλούμε την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στι γραμμές ε, δηλαδή και ειδικότερα στην διατροπική ανταγωνιστικότητα ανάμεσα δηλαδή στους διαφορετικούς τρόπους μεταφορών και να παρακολουθήσει το πώ ακριβώ εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη αυτή η ανταγωνιστικότητα. Αυτά από την πλευρά μα, κύριε Πρόεδρε, και είμαστε στη διάθεση των βουλευτών για να απαντήσουμε ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Έριξ, μα τάραξαν κάπω όλα αυτά βέβαια. Ο κ. Βαντενκάμπ έχει το λόγο. Βίμ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδιστή. αλλά πρέπει να πω ότι εσείς ε, πρόεδρε ήσασταν πολύ γρήγορος και ήταν προβληματικό να σας παρακολουθήσω. Θα συνεχίσω λοιπόν στα Ολλανδικά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως προανέφερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συχνά είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έχουμε υπέροχες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά έχουμε μια πολύ αρνητική επισκόπηση από το ελεκτικό συνέδριο. Και ευχαριστώ το Ελεκτικό συνέδριο γι' αυτό, διότι μας βοηθά στη δουλειά που κάνουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις λοιπόν. Από ό,τι κατάλαβα, οι διαδρομές, οι, διάδρομοι ε, του τέντη είναι και για τις γραμμές υψηλής ταχύτητας. Τελικά αυτό νόμιζα, αλλά φαίνεται δεν ισχύει. Αν είσαι σε ένα διάδρομο τέντη, θεωρούσα ότι σαν γραμμή υψηλής ταχύτητας ε, γίνεσαι αποδεκτή. Αλλά τελικά, ακούγοντάς σας, κύριε Ρίξ, συνεπέρανα ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείε από αυτού. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε, σα παρακαλώ. Δεύτερη ερώτηση. Η συμμετοχή των εθνικών αρχών. Οι διάδρομοι λοιπόν του TNT δεν ακολουθούνται πάντοτε από τις εθνικές αρχές ή δεν, τους, δεν, δεν γίνονται αποδεκτοί από αυτές τις αρχές. Αυτό είναι παράξενο διότι επενδύουμε δισεκατομμύρια για τα TNT και αν οι εθνικές αρχές ε, δεν ικανοποιούνται ε, και δεν τους αρέσουν, αυτό θα είναι πρόβλημα για μας. Τρίτον, κάτι που αναφέρεται στην έκθεση. Είπατε ότι δεν είναι πάντα αναγκαίο να ε, τοποθετείτε γραμμή υψηλής ταχύτητας διότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο αναβάθμισης υφισταμένων γραμμών. Δηλαδή αυτά τι είναι προγράμματα και έργα κυρούς τα, οι γραμμέ ψηλής ταχύτητα. Διότι θα πρέπει να τα κυρώσει αυτά τα έργα αν περί αυτού πρόκειται, αν είναι απλώς έργα κύρου και προβολής. Μετά, τέταρτον, είναι πολύ σύγχρονο να εισακούγονται όλοι. Ε, αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις όμως τελικά στην εκτέλεση έργων. Μήπως η συνεισφορά των πολιτών θα μπορούσε να είναι δομημένη, λίγο πιο καλά δομημένη. Πώς να το πω, να, να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο σαν ένα είδος καρτέλ. Οι Κινέζοι είναι διαφορετικοί ε, όσον αφορά την προσέγγιση τους, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικοί όσον αφορά την ε, κατάσταση ιδεοδρομικών ε, γραμμών υψηλής ταχύτητας και τη δρομολόγηση τρένων υψηλής ταχύτητας. έχουμε 11.000 εθνικούς κανονισμούς. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τι έχετε κάνει εσείς κύριε Ρίκε τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό για τους ρυθμιστικούς φορείς. Το ERA, η αρχή των σιδηροδρόμων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων δεν θα έπρεπε να μπορέσει να δώσει κάποιους προσανατολισμούς Ας βάλω και εγώ το δικό μου κερασάκι στην τούρτα μου. Η αγορά τρένων υψηλή ταχύτητα στη Γαλλία. Δεν νομίζω ότι αυτή η αγορά έχει ανοίξει και πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Αντιθέτω, παραμένει κλειστή στη Γαλλία. Παρα... Κρατούν του άλλου έξω. Αν δείτε το τέταρτο συνδρομικό πακέτο, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. δεν έπρεπε να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Eh, eh, eh, Ευχαριστώ. Είχαμε την ε, δυνατότητα να συζητήσουμε ήδη αυτή την, ε, τη σχετική γνωμοδότηση και γενικά θέλω να σας πω ότι δεν ε, συμφωνώ Υπάρχει μία αντίστοιχη έκθεση που είχε κάνει ένα άλλο ε, εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου, Αυστριακό και είχε φτάσει σε άλλα συμπεράσματα. Μην ξεχνάτε ότι στο μεταξύ υπήρξε η Συμφωνία του Παρισιού. Προσπαθούμε να φτιάξουμε συνδροδρομικά διευρωπαϊκά δίκτυα και για επιβάτες και για εμπορεύματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή μια αντίστοιχη ας πούμε κυκλοφορία με το αυτοκίνητο δεν είναι εφικτή. Είναι πάρα πολύ αντιφατική η έκθεσή σας. Από τη σκοπιά που εξετάζετε τα πράγματα, τα τρένα υψηλής ταχύτητας δεν είναι τόσο αποδοτικά, ε, δεν είναι τόσο όσο τα αεροδρόμια τουλάχιστον. Ε, Νομίζω ότι έχετε όμως προκατάληψη εναντίον των τρένων υψηλής ταχύτητας, ε, κύριε Χέντριξ. Αλλά και γενικά το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, όταν μας μιλάει για προβλήματα για τις διπλές γραμμές. Ε, δηλαδή τρένα υψηλή ταχύτητα και κανονικά τρένα. Λε και είναι πρόβλημα αυτό. Ή μιλάτε, α πούμε, για την ε, περιοχή που εξυπηρετείτε. 15-20 λεπτά, α πούμε, για να φτάσει σε αυτή την περιοχή με το αυτοκίνητο κα, κανεί. Ε, μπορεί να πάρει λέει, από 15-20 λεπτά μέχρι μία ώρα. Δεν ξέρω πώ κάνατε αυτή τη μελέτη. Δεν ξέρω με τι στοιχεία. Τι στοιχεία χρησιμοποίησατε. Επίσης, λέτε ότι κοστίζουν 395 εκατομμύρια ευρώ αυτές οι γραμμές. Τι είναι αυτό, όλα τα σχέδια, όλα αυτά τα έργα, ας πούμε, κοστίζουν τόσο. Η γραμμή τους δηλαδή, φαντάζομαι ένα χιλιόμετρο εννοείται. Επίσης, όταν μιλάτε για τους α, πολλαπλούς κανόνες θα ήθελα να ξέρω αν το 2018 το ελεκτικό συνέδριο έλαβε υπόψη το τέταρτο συνδρομικό πακέτο το οποίο συζήτησε και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για... Μιλάμε για την απλούστευση, ούτω ώστε να επιτρέψουμε να υπάρχει διασύνδεση μέσω τρένων ε, από μια χώρα στην άλλη. Δηλαδή να υπάρχει το πέρασμα ε, στα σύνορα. Η κυρία Γιούτο. Αντί, δεν θέλω να κάνω μία ερώτηση, θέλω να κάνω κάποιου προβληματισμού ακούσαμε, εκτός και αν κατάλαβα λάθος. Μα αποδείξατε με νούμερα μάλιστα ότι δεν χρειάζονται πάντα τρένα υψηλή ταχύτητα. και ότι από τις μελέτες και την ανάλυση που έγινε στα τα περασμένα χρόνια για το πώς σχεδιάστηκαν τα δίκτυα, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τα TEN-T δηλαδή, όταν ε, καθορίστηκαν ως γραμμές υψηλής ταχύτητας, ε, αυτές οι μελέτες λέτε ότι θα πρέπει να ξαναγίνουν, θα πρέπει να τις ξαναδούμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Γιατί αν ε, ο αριθμός των επιβατών που χρησιμοποιούν αυτές τις γραμμές είναι το 50% αυτού που προβλεπόταν και λιγότερο από το 50%, μιλάμε για χρήση πολύ κάτω από τις προσδοκίες. Επομένως, οι τρομερά δαπανηρές αυτές επενδύσεις που έγιναν και που θα γίνουν και στο μέλλον, θα πρέπει να δικαιολογούνται από, την, από μια ανάλυση κόστους-οφέλους. Συγκεκριμένη ανάλυση, ρεαλιστική ανάλυση, ούτως ώστε αυτά, αυτές οι επενδύσεις ήταν υπέρ των πολιτών. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε απέναντι στου πολίτε ότι για να κερδίσουμε ας πούμε, ένα λεπτό ας πούμε, θα πρέπει να ξοδέψουμε 90 εκατομμύρια ευρώ. Για να κερδίσουμε ένα λεπτό ταξιδιού. Έτσι, είμαστε γελοί τότε. Δεν ξέρω πώ θα δικαιολογήσω αυτό απέναντι στου πολίτε. Ότι πρέπει να ξοδεύουμε όλα αυτά τα λεφτά για να κερδίσουμε τι, ένα λεπτό. Να έχουμε ένα λεπτό ταξιδιού λιγότερο. Επομένω, το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε. Τι άλλες μελέτες προτείνετε ούτως ώστε να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε πορεία σε ό,τι αφορά τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Αν, υπά... αν αυτή η μελέτη και άλλες ενδεχομένως που έγιναν ή που θα γίνουν μπορεί να οδηγήσουν σε μια συνολική αναθεώρηση ενδεχομένως. Ε, θυμάμαι ότι η Επίτροπος μου ε, πριν από λίγους μήνες όταν μιλούσε για το τρίτο πακέτο για την κινητικότητα, μίλησε για το ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη να ληφθούν υπόψη όλα τα νέα στοιχεία και νέε απαιτήσει που συνδέονται με τα δίκτυα. Νέε αξιολογήσει ενδεχομένω, πιο επίκαιρε, για να τροποποιήσουμε ενδεχομένω την προσέγγιση μα. Την προσέγγιση για αυτέ τι επενδύσει. Επομένω, κάνατε αυτή την ανάλυση. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ έχω μια ερώτηση και κάποιες σκέψεις. Είμαι από το Φριούλι Βενέτσια Τζούλια και θέλουμε να έχουμε τη γραμμή ταιριέ στη Βενετία με γρήγορο τρένο. Αλλά είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Θέλω να πω ότι ο πληθυσμός της περιοχής μου αισθάνεται ότι έχει αποκλειστεί κάπως από το ολοκύκλωμα ενός εθνικού δικτύου τρένων υψηλή ταχύτητα και δημιουργείται και μια διακοπή, θα λέγαμε, τη ροή. Διότι εκεί που δεν υπάρχει τρένο υψηλή ταχύτητα υπάρχουν διαφορετικά τρένα. Οπότε στη Βενετία γίνεται η διακοπή αυτή τη ε, διαδρομή και αποτελεί ένα εμπόδιο όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου. Να προσθέσω ότι είναι και μια δυσυνοριακή περιοχή, οπότε η ερώτηση είναι τι συνέπειες υπάρχουν. Έχουμε οικονομικό όφελος. Μετά όμως είναι ποιο είναι το μειονέκτημα που μπορεί να υπάρχει όσον αφορά τη διασύνδεση και της έλλειψη, την έλλειψη των διασυνδέσεων, των links. Όταν υπάρχει μια διασύνδεση με το αεροπορική. Υπάρχει ανταγωνισμός με τον υψηλής ταχύτητας. Πρέπει να κάνουμε αξιολογήσεις ε, πάνω σε αυτό. Αν μιλάμε πάντα για τις δημόσιες μεταφορές, ε, υπάρχει και κανόνες παροχής υπηρεσίας περισσότερο παρά να εξετάζονται πτυχές αποκλειστικά εμπορικές και οικονομικές. Είναι δυνατόν κατά την άποψή σα, λαμβάνοντα υπόψη ότι είναι κάτι πολύ αφηρημένο να λάβουμε υπόψη εν γέννη τα ωφέλη, τα περιβαλλοντικά διότι αν έχουμε αποτελεσματική υπηρεσία που δίνουμε από πλευρά τρένων υψηλή ταχύτητα, δίνουμε και τη δυνατότητα μειώσεω των ε, εκπομπών που γίνονται όταν έχουμε μια σιδηροδρομική ε, διασύνδεση αντί να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα για τη διαδρομή αυτή. Κατά την άποψή μου, αυτή η μείωση των επιβατών ίσως εν μέρη να οφείλεται όχι στο ότι δεν είναι κατελκυστικό αλλά ότι υπάρχει κάποια οικονομική κρίση. Και ε, μια τέτοια υπηρεσία ε, για πολλούς έχει γίνει υψηλού επίπεδου το ΣΥΠΗΝ σε σχέση με την τοπική, τις τοπικές ε, μαζικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα κλείσω μέσω προσωπικών σκέψεων που θα εκφράσω. Το πρώτο σχόλιο που ακούστηκε. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των προδιαγραφών. Έχει δρομολογηθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ιδρομικών Μεταφορών. Λοιπόν, με τη συλλογή στοιχείων. Και έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα μείωση των κανόνων και των διατάξεων που είναι στον αριθμό 11.000. Άρα προχωρούμε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη. Λεπτομέρειες όσον αφορά τον απολογισμό άνθρακα, το γενικό. Δεν αναφέρει ένα θέμα το λεκτικό συνέδριο, που είναι η απόσβεση των επενδύσεων. η απόσβεση των επενδύσεων για τις υποδομές. Πόσο χρόνο χρειάζεται. Πότε θα υπάρξει κέρδος από τις επενδύσεις. Αν η διάρκεια απόσβεσης είναι πολύ μακρά και έχουμε διαφορετικές αποδόσεις, αυτό είναι κάτι που βαρύνει όσον αφορά την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας. Οι αναλύσεις σας για το κόστος γίνονται για κάθε έτος ή λαμβάνουν υπόψη το μακροπρόθεσμο θέμα των αποσβέσεων, το κόστος της ενέργειας και άλλα θέματα. Τρίτον, υπάρχουν και διεθνείς διασυνδέσεις όσον αφορά τα τρένα υψηλή ταχύτητας που ήταν πάρα, πάρα πολύ επιτυχής. Με το Θαλής, ποια είναι η άποψη το Θαλής. Μια κοινοπραξία όπως είναι το Θαλής, μια εταιρεία όπως το Θαλής, το Eurostar, που είναι εμπορική επιτυχία, αλλά είναι και δημοφιλή αυτά τα τρένα, αν κρίνουμε από την χρήση και από τη χρήση που κάνω και εγώ προσωπικά. Είδατε και το μέσο, τρένο ένα μέση υψηλή ταχύτητα, όπω την αποκαλώ. Σε κάποια τμήματα τη διαδρομή να τρέχει το τρένο με πάνω από 200 χιλιόμετρα, χωρί να ξεπερνάει όμω τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Έχετε κάποια άποψη όσον αφορά το θέμα της απόσβεσης των επενδύσεων του κόστους λειτουργίας κλπ. Ευχαριστώ όμως που ε, μας ε, εκθέσατε το θέμα. Πρέπει να κάνουμε βελτιώσεις κι εμείς. Χρειάζεται η γενική διοργάνωση να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και βλέπουμε ότι οι μεγάλες επιτυχίες είναι σε διεθνές επίπεδο που ξεκινάνε από Γαλλία, από Βρετανία, από Γερμανία. Η Ισπανία είναι λίγο θύμα, θα έλεγα, της διέλευσης των Πυρηναίων. Κάτι πρέπει να βελτιωθεί εκεί. Αλλά θα καταλήξουμε κάπου και εκεί. Έχετε πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι συνάδελφοι και βουλευτές. Ε, πολλά τα ερωτήματα που θέσατε θα προσπαθήσω να τα απαντήσω καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως, ε, όπως είπε βέβαια και ο κύριος Βαντεκάμπ, ε, πολλά από αυτά τα ερωτήματα απευθύνθηκαν και προς την Επιτροπή. Θα δώσουμε, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρόιτερ μετά. Okay, okay. Ja, äh, darf ich σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των ε, ε, διαδρόμων θα τα αφήσω στο συνάδελφο να τα απαντήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχολείο σας, σε ό,τι αφορά τον ε, ρόλο των εθνικών αρχών και το ότι δεν γίνεται δεκτή ε, η χρήση εδώ των ε, ε, διαδρόμων. Πραγματικά είναι περίεργο αυτό γιατί έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει, να λάβει μάλλον περισσότερε εκτελεστικέ εξουσίε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέου διαδρόμου. Όχι, θέλουμε απλά τα όσα προβλέπονται μέσα στον κανονισμό κατά την ευρωπαϊκά δίκτυα, όσα προβλέπονται μέσα στο μηχανισμό συνδέοντα τη Ευρώπη, να εφαρμοστούν στην πράξη. Εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν εθνικά έργα, εκεί λειτουργούν και ε, καλά οι ε, γραμμές υψηλής ταχύτητας. Τα προβλήματα τα εντοπίζουμε ακριβώς στις διασυνοριακές συνδέσεις, στις διασυνοριακές γραμμές και γι' αυτό λοιπόν δώσαμε προτεραιότητα σε αυτό το τομέα. Γιατί εκεί βλέπουμε να υπάρχουν ε, προβλήματα εκεί υπάρχουν ελλείψεις και εκεί θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων. Ναι, υπάρχουν και κάποια project τα οποία πραγματικά έχουν ρόλο ιδιαίτερου κύρου πρεστή. Ε, στην ε, παράγραφο 46 της έκθεσης ε, και υπάρχει και ένας πίνακας που αναφέρεται για παράδειγμα στη σύνδεση μεταξύ Βενετίας και τρέστη. Δηλαδή εκεί τι λέμε, ότι με αυτήν την διαφορά είπαμε τον... 10 λεπτών σε ό,τι αφορά το χρόνο του ταξιδίου υπάρχει εξοικονόμηση 570 εκατομμυρίων ε, ευρώ. Ε, και αναφέραμε επίση ότι, για παράδειγμα, στη Γερμανία και στη Γαλλία θα πρέπει να γίνει μια ανα, ε, αναθεώρηση, μια επανεξέταση του κατά πόσο οι ανάγκε για την χρήση αυτών των γραμμών υψηλή ταχύτητα παραμένει. Γιατί βέβαια έχουν γίνει σημαντικέ επενδύσει σε αυτέ τι δύο χώρε και θα πρέπει να, είναι, να διασφαλίζεται ότι υπάρχει κατάλληλη αξιοποίηση των επενδύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη του περιορισμού, αν θέλετε, των δικαιωμάτων των επιβατών σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή του, νομίζω πω εδώ δεν θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εμά, αλλά στα εθνικά κράτη-μέλη. Φυσικά οι διαδικασίε σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο χρειάζονται κάποιο χρόνο να εκτελεστούν, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε και, τις, ε, και τη θετική πλευρά σε ό,τι αφορά δηλαδή την συνεισφορά των ε, πολιτών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την πρόληψη από, ένα από μια σειρά από διαφορετικά είδη μόλυνση. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Δηλαδή, θα πρέπει να πληρώνουν ορισμένε προποθέσει και οι κατασκευαστέ και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρξει τήρηση των σχετικών ε, προποθέσεων. Και εδώ παίζει βέβαια ρόλο και η ύπαρξη one-stop shop, δηλαδή ε, θεωρείται μια εξυπηρέτηση, σημείων μια εξυπηρέτηση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα διασυνοριακά έργα. και το σχετικό έργο το οποίο κατασκευάζεται τώρα με τα τούνελ είναι πάρα πολύ σημαντικό από τα μεγαλύτερα ανά τον κόσμο, αλλά βλέπουμε ότι άλλες είναι διαδικασίες που τρέχουν στην Ιταλία και άλλες ε, στην Αυστρία και εδώ θα πρέπει να κάνουμε ε, κάποια προσπάθεια για περισσότερη εναρμόνιση. Σε ό,τι αφορά ε, τι διατάξει, 11.000 διατάξει που είπαμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν στο εθνικό επίπεδο, θα, θα δώσω το λόγο στον συναδέλφο, αλλά εδώ επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε με διατάξει εθνικέ. Γιατί αναφέρθηκε ξανά και ξανά το τέταρτο πακέτο για του σιδηροδρόμου. Μα σα λέω ότι αυτέ οι διατάξει 11.000 είναι εθνικού χαρακτήρα που καθιστούν τόσο δύσκολη τη διαλειτουργικότητα. Και ο συνάδελφος θα αναφερθεί και περαιτέρω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων και του σχετικού ε, κινδύνους, ε, στην ε, παράγραφο 87 αναφέρομαστε σε αυτούς, για παράδειγμα, τις πολύ μεγάλες προθεσμίες, για παράδειγμα, δεκαετής καθυστερήσεις, οι δυνατότητες δεκαετούς καθυστέρησης και ούτω καθεξής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο πραγματικός ανταγωνισμός, για παράδειγμα, σε αυτές τις γραμμές θα ξεκινήσει το 2035. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πακέτο έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένε εξαιρέσει για συγκεκριμένε επιχειρήσει, συγκεκριμένου ε, operators και βέβαια σε σχέση με αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο γιατί εδώ ε, έχουμε να κάνουμε με ισχύουσα νομοθεσία. Απλώ λέμε ότι μπορεί να υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο. Ε, σε ό,τι αφορά κάποιες αμφιβολίες οι οποίες αναφέρθηκαν στη σχετική εκθέση του ελεκτικού συνεδρίου. το, η δική μας υποχρέωση είναι να προβλέπουμε ε, και να προβαίνουμε σε, μια, σε ένα διπλό έλεγχο. Και πάντοτε γίνεται μια αξιολόγηση θετικών και αρνητικών αντικτύπων και στο πλαίσιο αυτό ε, πάντοτε συμβουλευόμαστε τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ε, και με βάση τις δικές τους μελέτες κινούμα, κινούμαστε περαιτέρω και το ίδιο κάναμε και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, με κατηγορήσατε ότι είμαι πολύ αρνητικός στην αξιολόγησή μου. Όχι, δεν συμφωνώ. Ε, σας ε, παραπέμπω εδώ στην πρώτη παράγραφο της σύνοψης της έκθεσής μας ε, και σας τη διαβάζω στα αγγλικά. Ε, ο σιδηρόδρομο αποτελεί ένα ασφαλή, ε, φιλοπεριβαλλοντικό, αποτελεσματικό τρόπο, ο οποίος ε, μπορεί να υποστηρίξει τις, τους στόχους της πολιτικής συνοχής και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι αρμόδιος για όλη αυτή την έκθεση και είμαι αρμόδιος και για την πρώτη παράγραφο. Άρα λοιπόν το αναφέρουμε αυτό το στοιχείο στην πρώτη παράγραφο, αλλά και στο τέλος της έκθεσης υπάρχει μια την παραβολή όχι μόνο μεταξύ σιδηροδρόμων και για παράδειγμα αέριων ε, και οδικών μεταφορών, αλλά έχουμε κάνει και πιο αναλυτική ε, εξέταση σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες συνδέσεις ε, έναντι για παράδειγμα των αέριων μεταφορών. Από την πλευρά δηλαδή πάντων των γραμμών υψηλής ταχύτητας. Και επίσης σε όλα αυτά τα τέσσερα διασυνοριακά έργα στα οποία αναφερόμαστε, ε, στα οποία ακριβώς το ζητούμενο είναι να επιτύχουμε προστιθέμενη αξία, δηλαδή υψηλότερη αξία από την εθνική. Σε αυτά λοιπόν τα τέσσερα διασυνοριακά έργα ε, υπήρξαν πολύ σημαντικές δυσκολίες τις οποίες διαπιστώσαμε. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν υπάρχει δίκτυο ευρωπαϊκό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέρη ενός δικτύου τα οποία συνθέτουν ένα όλο, ένα συνολικό δίκτυο και γι' αυτό ακριβώς δικαιολογείται ο τίτλος που δώσαμε στην έκθεσή μας. Επίσης είπατε αυτά τα 69 ε, δις ευρώ ανά ε, λεπτό που γλιτώνουμε σε ό,τι αφορά την ε, το, το χρόνο ταξιδίου, η μέση ε, αξία είναι 90 εκατομμύρια εξοικονόμησης. Και σε ό,τι αφορά την σύνδεση μόναχο του Τκάρδης, εκεί έχουμε την, το, το μέγιστο ποσό 369 εκατομμύρια ευρώ. Κατά μέσο όρο 90 εκατομμύρια ευρώ είναι εκείνα τα οποία επενδύονται για να επιτύχουμε ένα λεπτό λιγότερου χρόνου ταξιδίου. Άρα λοιπόν κάναμε μια σωστή ε, παραβολή των σχετικών ε, δεδομένων και είδαμε τι ακριβώ εξοικονομούμε σε επίπεδο υψηλή ταχύτητα σε ε, σύγκριση με συμβατική ταχύτητα. Γιατί θέλουμε λοιπόν να έχουμε και διαφανή δεδομένα, γιατί δεν θέλουμε απλώ και μόνο αριθμού, θέλουμε και συγκεκριμένε συγκρίσει. Επίση, ε, αναφερθήκατε και συνάδελφε στην, ε, ε, ε, κυρία στι 11.000 διατάξει, τι οποίε όπω σα είπα θα αναφερθεί ο συνάδελφό μου. Επίση, τέθηκε το ζήτημα του κατά πόσο τελικά δικαιολογούνται είναι οι επενδύσει που έχουν γίνει ή όχι. Εντάξει, δεν νομίζω πω θέσατε ένα ερώτημα, απλώ ε, ασκήσατε μια κριτική. Πάντω, εκείνο που εμεί διαπιστώνουμε ε, και το οποίο αποτελεί μια έλλειψη είναι το γεγονό ότι δεν έχουμε συστημική χρήση, συστηματική μάλλον συγγνώμη, χρήση αναλύσεων κόστο αποτελέσματο. Ε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιε αναλύσει μετά από τη λήψη τη σχετική απόφαση σε ό,τι αφορά το τούνελ Μπρένερ του 2007 Ε, και έκτοτε βέβαια έχουν, γίνει, έχουν συμβεί πολλά. Το, τα πάνε σχετικά αυξήθηκαν το χρονοδιάγραμμα ε, μεγάλωσε αλλά οι εκτιμήσει σε ό,τι αφορά τι αναμενόμενες ε, συνδρομικές μεταφορές φορτίων μειώθηκαν οπότε πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή αξιολόγηση κόστους αποτελέσματος γιατί πάντοτε χρειαζόμαστε στοιχεία για να διαπιστώνουμε κατά πόσο έχει νόημα να γίνει μια επένδυση ή αντιθέτω δεν έχει νόημα μια άλλη επένδυση και ε, υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν όπω έγινε όπω σα είπα στη σύνδεση μεταξύ ε, και Βενετία, όπου μπορούν καλύτερα να αξιοποιηθούν τα ε, κονδύλια. Και αντιμόντα αναφερθήκατε τώρα στην ε, ίδια αυτή τη γραμμή βενετία σε Τρίστη και εδώ σα παραπέμπω στον πίνακα 3 μετά από την παράγραφο 46 της έκθεσής μας. Ναι, δεν ξέρω ποια θα ήταν τα μειονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν από, μια τέτοια αναβάθμιση, αλλά πάντως και στην ενότητα εκείνη στην οποία αναφερόμαστε στην, στην αυξημένη αξία για του ε, επιβάτες λέμε ότι για εκείνες τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συνδέσεις ε, πολύ σπάνια σταματάνε σχετικά τρένα και σε αυτές τις ε, περιοχές σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή στη συγκεκριμένη σύνδεση, τα πράγματα έχουν λειτουργήσει καλύτερα, αλλά γενικά αυτό δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, δηλαδή αυτή η σύνδεση αυτών των περιοχών. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τι ενεργέ κυκλοφορίε και την αλληλεπικάλυψη των ίδιων δηλαδή διαδρομών με του σιδηρόδρομου. Πράγματι, ρίξαμε μια ματιά Ε, στην Ιαπωνία με, με τις αλληλεπικαλύψεις που υπάρχουν εκεί γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε μία ε, σύγκριση. και μιλάμε εδώ βέβαια για τελείως διαφορετικά, ε, διαφορετικές ανάγκες σε επίπεδο μετακίνησης επιβατών στις 163 εκατομμυρίων σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ενδύσεις μεταξύ πολύ μεγάλων πόλεων. Και οι συγκρίσει του κόστου εδώ ε, που βέβαια κάνουμε δείχνουν ότι τα νούμερα δεν είναι πολύ διαφορετικά σε ό,τι αφορά το κόστο. Οπότε πάντοτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και αυτή τη διάσταση τη χρήση δηλαδή των ε, δικτύων. Και έρχομαι, σε αυτό, έρχομαι εδώ σε αυτό που ανέφερε και ο Πρόεδρο. Δηλαδή πάντοτε θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη η κατασκευή ε, τέτοιων ε, γραμμών ε, σιδηροδρόμων ή σιδηροδρόμων υψηλή ταχύτητα. Εκείνο που λέμε εμεί πάντοτε είναι ότι θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση του κατά πόσο έχει νόημα, είναι αποτελεσματική, έχει σωστή σχέση κόστου αποτελέσματο σε μια γραμμή ή αν αντιθέτω υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν όπω έγινε, όπω σα είπα, στην Ιταλία, όπω έχει γίνει στη Γερμανία. Ε, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει σε αυτά τα μεγάλα έργα έχουμε τόσο μεγάλου ε, ε, χρονικού ορίζοντε κατασκευή, έτσι ώστε οι αρχικέ εκτιμήσει να μην ισχύουν και εκεί θα πρέπει να γίνεται μια νέα αξιολόγηση. Γιατί βέβαια ο στόχο πάντοτε είναι να καλύπτονται οι φυστάμενε ανάγκε. Δεν είναι αυτό ο σκοπό η δημιουργία τέτοιων γραμμών. Ο σκοπό είναι να καλύψουμε με αποτελεσματικό τρόπο ε, τι ε, ανάγκε των πολιτών. Προφανώ από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τι γραμμέ τι οποίε εξετάσαμε και πρέπει προφανώ να λάβουμε υπόψη μα το αν έχουμε μεταφορέ επιβατών ή φορτίων. Σε, σε αυτέ τι τρει γραμμέ που ελέγξαμε, σε εκείνη την περίπτωση είχαμε, ε, βρισκόμασταν κάτω από το στόχο των 9 εκατομμυρίων. Οπότε τα πρέπει, όπω είπα, πάντοτε να γίνουν αυτέ οι αξιολογήσει. Και έρχομαι τώρα στα όσα είπε και ο πρόεδρο, ο οποίο αναφέρθηκε στη διαλειτουργικότητα και ε, στι εργασίε ΕΡΑ. Και εδώ και πάλι θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, την. να βλέπουμε κατά πόσο έχουν πραγματικά ε, Μπορούσαμε να κερδίσουμε και πάλι από τις επενδύσεις μας ε, με τις, ε, τα σχετικά κονδύλια. Να πούμε ότι ε, δυστυχώς δεν έγινε η σχετική εκτίμηση σε ό,τι αφορά τους αεροδρόμους. Το κάναμε σε ό,τι αφορά τις αέρες κυκλοφορίας, αλλά όχι σε σχέση με τις οδρομικές γραμμές. Εξετάσαμε τα αστικά κέντρα, εξετάσαμε τις, τα benchmarking, δηλαδή τις συγκριτικές μελέτες, αλλά δεν κάναμε μια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τις αποσβέσεις των σχετικών επενδύσεων, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις, ε, τα θετικά παραδείγματα, ε, πράγματι έχετε δίκιο. Το Eurostar πραγματικά αποτελεί ένα παράδειγμα ως προς τα όσα έχουμε. Βέβαια γνωρίζουμε τα προβλήματα που είχαν προκύψει και τότε βέβαια έχουν ε, βελτιωθεί και αυτή την περίοδο λειτουργεί σωστά εν λόγω γραμμή. Απλώς εμείς εδώ αναφερόμαστε και σε, προφανώς και σε επιτυχημένες γραμμές ε, στη Βαρκελόνη, ε, στο, στο Παρίσι, ε, σύνδεση μεταξύ Ρώμης και Τουρίνου, όπου έχουμε πραγματικά και υψηλό αριθμό επιβατών, όπου έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες και καλά αποτελέσματα. Χωρίς να γνωρίσουμε επακριβώς όλα τα στοιχεία. Δηλαδή υπάρχουν και επιτυχημένα project φυσικά. Υπάρχουν και, εκεί θα πρέπει να βλέπουμε ποιε είναι οι συνθήκε υπό τι οποίε υλοποιούνται και τρέχουν αυτά τα έργα, για να τα συγκρίνουμε ακριβώ με εκείνα τα έργα που δεν λειτουργούν καλά. Και εδώ επανερχόμαστε ακριβώ στο ίδιο ε, στοιχείο που αναφέραμε, ότι δεν λαμβάνονται καταλήλω υπόψη ασιατικά σχετικά στοιχεία, δεν υπάρχει αξιολόγηση ε, κόστου αποτελέσματο, ε, δεν λαμβάνονται υπόψη ανάγκε των ε, πολιτών εκεί και οι σχετικοί σταθμοί, για παράδειγμα. Δηλαδή, Ε, με όλες τις ε, στάσεις για παράδειγμα ε, σε κάθε στάση μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ενός μια διαδρομή διαδρομής κατά έως 16 λεπτά και μειώνεται και ο σχετικός χρόνος ταχύτητας, η σχετική ταχύτητα του τρένου οπότε θα πρέπει πάντοτε να αξιολογούμε και πού ακριβώς και ποιες είναι οι στάσεις οι οποίες γίνονται. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα τη ταχύτητα, της ταχύτητας γενικά στην οποία αναφερθήκατε στον παράδειγμα 5 για όποιον ενδιαφέρεται αναφέρουμε τη μέση ταχύτητα των ε, διαφορετικών γραμμών. Και τα θετικά παραδείγματα και τα λιγότερο θετικά. Ε, ποια είναι δηλαδή η μέση ταχύτητα, ε, ποια είναι η ανώτατη δυνατότητα. Και για παράδειγμα ανάμεσα σε Μαδρίτη και Βαρκελόνη φτάνουμε πάνω από τα 200 χιλιόμετρα ω μέση ταχύτητα. Γιατί προφανώ εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει, πρέπει να δίνει το τρένο και ούτω καθεξή. Αλλά πάντοτε κάνουμε συγκριτικέ μελέτε αλλά υπάρχουν γραμμές οι οποίες φτάνουν στο 70-80% της αξιοποίησης της μέγιστης ταχύτητάς τους, αλλά διαπιστώνουμε εδώ λοιπόν στις ε, γραμμές ε, που κάναμε, ε, στις, στις που εξετάσαμε ότι βρισκόμαστε πολύ πολύ χαμηλά, δηλαδή κάτω από το ίμιση της ανώτατης αυτής ταχύτητας, πράγμα το οποίο δείχνει ακριβώς ότι δεν αξιοποιείται πλήρως εν λόγω επένδυση. Και αν μου επιτρέπετε, πρόεδρε, να δώσω τον επικεφαλής της ερμητικής μας ομάδας σε περαιτέρω διευκρινήσει. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε εδώ, σε αυτή την ακρόση. Εξετάσαμε τα ωράρια στα αεροδρόμια κλπ. πριν πω συγκεκριμένα θέματα. Επισήμως ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θετικότατη συνεργασία μαζί τους, πολύ επαγγελματική, η υλοποίηση του ελέγχου με διαφάνεια, χωρίς εκπλήξεις και από τις δύο πλευρές, όσον αφορά να ξεκαθαρίσουμε ότι όπως ανέφερε και ο κύριος Έριξ, έχουμε θετική αρχική προσέγγιση, θετικά μηνύματα, τα οποία όμως τελικά χάνονται στην πολιτική επικοινωνία που ακολουθούμε. Σημαντικό όμω να τονίζονται τα θετικά στοιχεία, γι' αυτό ξεκινάμε και από εκεί. Σας ζητώ λοιπόν να διαβάσετε προσεκτικά την έκθεση, τις λεπτομέρειες. Εκεί κρύβεται και ο διάβολος άλλωστε. Στι λεπτομέρειε. Άριστη συνεργασία μέχρι τέλους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη εισέπραξαν πολλές από τις συστάσεις μας, τις συμπεριέλαβαν στην ε, αναμενόμενη νομοθεσία, στο ΣΕΦ 2 ή την πρόταση συγχρονισμού ε, των διαφόρων πολιτικών έλαβαν υπόψη τις ε, παρατηρήσεις μας και τα σχολιά μας. πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις όσον αφορά επιδόσεις στο μέλλον. Ο κύριος Βάντερ Κάμπ έκανε ενδιαφέρουσε ερωτήσεις. Οι διάδρομοι TEN-T εμπλέκουν και τα κράτη-μέλη. Δεν θα έπρεπε να δεσμεύονται τα κράτη-μέλη από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Απάντηση είναι ναι. Θα έπρεπε, ασφαλώς. Κανείς δεν του ζήτησε να ζητήσουν τα χρήματα από τι Βρυξέλλε. Αν ζητούν χρήματα από τις Βρυξέλλε, πρέπει να μοιραζόμαστε και εμείς ένα κομμάτι από την εθνική κυριαρχία. Περί αυτού πρόκειται. Συζητήθηκε αυτό και στο Συμβούλιο. Θέσαμε προκλητική ερώτηση. Είναι σχέδιο ή πολιτικό στόχο, ήταν η ερώτηση. Αν ήταν ένα σχέδιο, αν συμφωνούν όλοι, πρέπει να εφαρμόζεται. Δηλαδή, μέχρι το 2030 θα πρέπει να τριπλασιαστεί το βασικό δίκτυο. Έχουμε στοιχεία όμω τελικά που δείχνουν δεν θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Γι' αυτό στην πρώτη σύσταση είπαμε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άρα να αναθεωρήσουμε το όλο πρόγραμμα για να γίνει ρεαλιστικό. Και εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπάρχουν για να είναι ρεαλιστική και υλοποίηση. Να έχουμε κινέζικες διαδικασίες ούτως πίν για να προχωρήσουμε. Συμφωνώ. Ίσως πρέπει να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση σε σχέση με την παρούσα σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να μπλοκάρουμε τις διαδικασίες για πολλούς λόγους, να μειώσουμε τη διάρκεια των, μάλλον να επιβραδύνουμε τις διαδικασίες και να χρειάζεται πολλής χρόνος. Και αυτή η πρόταση για ενιαία θηρίδα που κάναμε ίσως οδηγεί σε κάποιο εξυγχρονισμό και επιτάχυνση. Δεν ξέρω αν είχαμε, ε, θα έχουμε ακόμα 11.000 διατάξεις. Το 2018 έχουμε. Μας το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε 11.000 διατάξεις. Εάν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδεοδρόμου δεν κάνει τη δουλειά της, την κάνει. Αλλά δεν εργάζεται με πολύ ψηλή ταχύτητα. Ίσως είναι γενέ στοιχείο τη διαδικασίας, ότι είναι χρονοβόρα. Κάτι κάνει αυτή η υπηρεσία, ναι, κάνει. Συνομιλήσαμε, το κουβεντιάσαμε, μας δώσαν λεπτομέρειες όσον αφορά το τι κάνουν. Η πρόοδος γίνεται με πολύ αργό ρυθμό. Τι προτείναμε, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ε, για να ανοίξει η αγορά τη Γαλλία στον αφορά τα τρένα υψηλή ταχύτητα και στο τέταρτο πακέτο να έχουμε αλλαγέ πρόσφατα στη Γαλλία. Από όταν ανέλαβε νέο πρόεδρο ο κ. Μακρόν, κάτι προσπαθεί να κάνει. Όχι μόνο διότι το Εθνικό ελεκτικό Συνέδριο είπε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χρέος το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι τμήμα της διαδικασίας, χρειάζεται πολύς χρόνος, θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Εν τω μεταξύ, δαπανούμε πολλά χρήματα με μεγάλη ταχύτητα για τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Για το Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν γνώριζα για αυτή την έκθεση. Εγώ είμαι ο ελεγκτής. Ηγούμε του ελέγχου. Και στέλναμε ομάδες στην Αυστρία Στείλαμε κόσμο στη Γερμανία, στην Ιταλία και παίρνω πληροφορίες από τις ομάδες μου. Δεν έλαβα όμως αυτή την αυστριακή έκθεση. Κάνω τον έλεγχο όπως θα έπρεπε, μεθοδολογικά. Είχαμε στοιχεία. Και ότι δεν υπάρχει σχεδιασμό στη Γερμανία. Δεν προσπαθούν να επενδύσουν στον βόρειο άξονα προς τον Μπρένερ, ενώ κατασκευάζουν ήδη Αυστριακοί και νότιους άξονες προς την Ιταλία. Ξεκίνησαν κατασκευές. Έλλειψη επικοινωνίας, πώς να το πω, έλλειψη συντονισμού, να το πω, έλλειψη έγκαιρης υλοποίησης, ας το θέσουμε έτσι και από τις δύο πλευρές. Το ίδιο ισχύει για την Πορτογαλία. Και η Πορτογαλία δεν θα κατασκευάσει τις υδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας. Τουλάχιστον μέχρι λήξη του ελέγχου δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο. Τα ίδια στη χώρα των Βάσκων. Η Ισπανία κατασκευάζει στη χώρα των Βάσκων. Η Γαλλία δεν κάνει τα προβλεπόμενα να συνδεθεί το Μπορντό με το Ντάξ με τρένο υψηλής ταχύτητας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι συμβατικές γραμμές, αλλά το δίκτυο υψηλή ταχύτητα είναι που συζητούμε. Τέταρτο πακέτο των σιδηροδρόμων, το συζητήσαμε. Το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, λέμε κάτι αρνητικό, όχι. Έχουμε το παράρτημα 4. Εκεί ξεκαθαρίζουμε ότι στην Ισπανία κατά κεφαλή η χρηματοδότηση με Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ψηλότερη από τις άλλα Λογικό. Διότι οι Ισπανοί κατασκευάζουν εντελώς καινούριο δίκτυο. Βλέποντας δίκτες Επιβάτε ένα χιλιόμετρο, επιβάτες ανά χιλιόμετρο κεφαλή. Είναι πολύ χαμηλά τα στοιχεία, δεν είναι κάτι παράξενο. Είναι καινούριο το δίκτυο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ε, ετερόκλητα πράγματα. Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά το κόστος ελήψεως διασυνδέσεων. Καλή παρατήρηση, καλή. Κάναμε μελέτη σχετικά με αυτό στην υποσημείωση παριθμών 23. Αναφέρουμε τη μελέτη που έγινε το 2015. Τίτλος. Κόστος μη ολοκλήρωσης του ΤΕΝΤΗ». Υποσημείωση 23. Το αναφέρουμε και. Σωστά. Έπρεπε να έχουμε αποτέλεσμα δικτύου, χρήσης δικτύου. Όσο μας λείπουν οι κρίκοι, διασυνδέσεις και όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση του δικτύου, τόσο λιγότερο αποτελεσματικό είναι το δίκτυο. Καθυστερεί η αποτελεσματικό του δικτύου. Και αυτό είναι το βασικό θέμα. Υπάρχουν κάποια τμήματα του δικτύου που ίσως οικονομικά δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα για να κατασκευαστούν από ένα κάτω μέλος. Δεν υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος. Αν υπήρχε διασύνδεση όμως θα υπήρχε αποτέλεσμα λόγω δικτύου. Εδώ τίθεται το ζήτημα. Ενδιαφέρουσα η μελέτη που αναφέρεται στην υποσημείωση 23. Εξετάσαμε περιβολατικά στοιχεία. Στην υποσημείωση 17 της έκθεσης. Εκεί συμπεράναμε ότι εν γέννη είναι αποδεκτό ότι είναι πολύ εποφελής ε, η προσέγγιση αυτή για το περιβάλλον. Είχαμε κάποιες επιτυχίες λοιπόν σε αυτές τις γραμμές, αναφέραμε τις επιτυχίες, προσπαθήσαμε να έχουμε ένα σύστημα ε, στάθμισης, βαθμολόγησης, Παρίσι, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, πήραμε στοιχεία από Παρίσι, Βρυξέλλες, δεν πήραμε στοιχεία για το Βρυξέλλες, Άμστερνταμ. Ξέρουμε ότι κάποια τμήματα λειτουργούν σωστά, κάποια άλλα όχι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Τι προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε μέσω της εκθέσεως. Πρώτον, δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα για κάποιες γραμμές. Δεύτερον, δεν είμαστε πάντα σε θέση να αποσαφηνίσουμε ότι είναι κάτι πολύ καλό. Ε, οι αποφάσεις ελήφθησαν εμπεριστατωμένα ε, υπάρχει ανάλυση, έλλειψη ελ, ανάλυσης κόστους κόστους-οφέλους και κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε τι δεν αποδίδει ε, λόγω υποδομών ή λόγω υπηρεσιών. Όταν δεν έχουμε κάποιες υπηρεσίες, έχουμε γραμμές που είναι ανοιχτές για ανταγωνισμό, όπως στην Ιταλία. Περισσότερα τρένα υψηλότερε, καλύτερε υπηρεσίε, καλύτερε τιμέ για του επιβάτε. άλλα κράτη-μέλη δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Κρίμα. Διότι όλοι στι χώρε επενδύουμε. Αυτά και θα σταματήσω εδώ. Τι είναι αυτό. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή ε, που είναι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι έχει πράγματα να μας πει κάποιες, ε, προβληματισμούς. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν καλωσορίζει τη σημερινή έκθεση και τις συστάσεις του ελληνικού Συνεδρίου. Υποστηρίζουμε τους στόχους του Ελεκτικού Συνεδρίου που είναι να ξοδεύουμε σωστά τα λεφτά των φορολογουμένων. Όμως, είναι σημαντικό να διαβάσει κανείς ολόκληρη την έκθεση, όχι αποσπασματικά. Καταρχάς, να τονίσω ότι η Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη διαδικασία προγραμματισμού. Ο κανονισμός TEN-T ε, μας δίνει την μακροπρόθεσμη στρατηγική με προτεραιότητες ε, για ένα πλήρες δίκτυο και ημερομηνίε οδοκλήρωση του δικτύου μέχρι το 2030. Υπάρχει και μια νέα διαχείριση επίσης με αυτή την νομοθεσία, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διαχείριση σημαίνει βασικούς ε, διαδρόμους. Ευρωπαϊκοί συντονιστές θα διευκολύνουν την εφαρμογή και διασύνδεση με τα μέσα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το ΣΕΦ, το Connecting Europe Facility. Βεβαίως αυτά μπορούμε να τα βελτιώσουμε περαιτέρω και η Κομισιόν θέλει να βρει τα κατάλληλα μέτρα ούτω ώστε να δώσει συνέχεια στις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Αναφέρθηκε νέα πρόταση για το ΣΕΦ και η πρόταση απτούντευσης για τα έξυπνα TNT που έχει υποβληθεί από την Κομισιόν και θα ε, επιταχύνει την ολοκληρώση των διαδρόμων και του δικτύου TNT. Επίσης, δύο εκτελεστικές αποφάσεις έχουμε υιοθετήσει μέχρι στιγμή και ετοιμάζουμε άλλε δύο εκτελεστικές αποφάσεις. Αυτά είναι απάντηση στι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα απαντήσω σύντομα σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Ο ιτεπλασιασμός ε, των τρένων υψηλής ταχύτητας είναι δυνατός, αλλά χρειάζεται χρόνο. Αν δείτε τι έχει γίνει μέχρι το 2011 και μετά, και τι μπορεί να γίνει μέχρι το 2030, νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό ο στόχο του πλαισιασμού. Θα απαιτήσει όμω ε, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και όλοι οι ενδιαφερομένοι να συνεργαστούν. Ε, δεν πρέπει όλα να γίνουν επίση ε, με ταχύτητε 300 και, αλλά και το 200 και είναι μια ταχύτητα μέσω υψηλή, ας πούμε, που υπάρχει σε πολλές χώρες ε, συνοχής, παραδείγματος χάρη στην Πολωνία, 250 κτλ. Αλλά και πολλά έργα σε δυτικές χώρες που στοχεύουν σε αυτές τις ταχύτητες. Ας πούμε, ε, η σύνδεση Βιέννης και Νίκιας. Επίσης, ε, υπάρχει διασύνδεση με το τέταρτο πακέτο συντηροδρόμων για να εγκαταλείψουμε τους εθνικούς κανόνες. Και όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, ε, είναι κατάλληλη στιγμή, γιατί ο ΑΕΡΑ δουλεύει και ελπίζουμε οι πολλοί εθνικοί κανόνες και ποικίλοι και διάσπαρτοι που υπάρχουν μέχρι το 2019 να καταργηθούν. Τώρα, για κάποια διασυνοριακά έργα, μιλήσατε Πρόεδρε για την αποτελεσματικότητα του δικτύου υψηλής ταχύτητας μεταξύ Παρισιού, Βρυξελών, ε, Άμστερνταμ και Κολονίας. Είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασία ε, αυτών των τρένων ψηλή ταχύτητα. Ε, υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα με τη συνεργασία να εφαρμοστούν και άλλα. Ε, είναι δύσκολο και κοπιαστικό να γίνει, αλλά προσπαθούμε. Ε, το Brenner θα ολοκληρωθεί με το 2026 και υπάρχουν και άξονες ε, προσπέλασης που δημιουργούνται λίγο-λίγο. Η διασύνδεση μέσω των Άλπιων χρειάζεται μεγάλες σύραγγε, ούτω ώστε να υπάρχει εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα. Επίσης ε, και σε διασυνδέσεις με το Τωρίνο κτλ. Για τις, τη σύνδεση της Ισπανίας και Γαλλίας κτλ. στην Ιβυρική Χερσόνησο, τα τρία ενδιαφέροντα κράτη-μέλη συνεργάζονται ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν χτίζει μόνο το ένα κράτος και τα άλλα δρανούν, αλλά όλοι χτίζουν. Ε, και ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ε, τις συστάσεις επίσης ε, του Ελληνικού Συνεδρίου τις ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και ελπίζουμε μαζί με το Κοινοβούλιο, και, το Κοινοβούλιο καθώς και τις προτάσεις για το ΣΕΦ2 κτλ. θα δώσουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τώρα τους δύο ομιλητές από το Ελεκτικό Συνέδριο. Και τελείωσε το δικό σας το σημείο. Τελειώσαμε. Όχι, λέει ο κύριος Βάντεκάμπ. Καταλαβαίνω την αισιοδοξία, ε, αλλά δεν με καθησυχάσετε σε ό,τι αφορά τη Γερμανία και την Βαβαρία, σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση στον Μπρένερ. Δεν συμβαίνει τίποτα εκεί. Ε, πήγαμε τον κύριο Κράμερ εκεί πέρα εγώ και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι επισκεφτήκαμε τον Μπρένερ. Οι... οι Ιταλοί χτίζουν, οι Αυστριακοί χτίζουν. Α, ήσασταν κι εσεί πρόεδρε. Ναι. Κάναμε και ωραίες φωτογραφίε μάλιστα. Πήραμε πολύ ωραίες φωτογραφίε. Ε? Αλλά όμως οι Γερμανοί δεν κάνουν τίποτα καλό θα ήταν ο υπεύθυνο από το ελεγκτικό συνέδριο ή μάλλον της ε, Κομισιόν να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Κλείνω τη συζήτηση. Σας δώσαμε πολύ περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο. Κοιτάξτε, μπορούμε να συνεχίσουμε ατέρμον εδώ πέρα, να συζητάμε κάθε γραμμή. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Βεβαίω, ε, το Brenner είναι το πιο θεαματικό γιατί είναι το μεγαλύτερο εργοτάξιο αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό να εστιάσουμε ξανά σε μια τέτοια συζήτηση ε, για να δούμε κατά πόσο προχωράνε αυτά τα έργα. Υπάρχει συνέπεια, ας πούμε, και στο διοσυναριακό επίπεδο κτλ. Σε... Θα ξανακαλέσουμε βέβαια στο ελεγκτικό συνέδριο για να μας κάνει παρουσίαση. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για μεγάλα έργα, πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πολύ ωραία. Και τώρα θα μιλήσουμε για, την, ε, για το μηχανισμό για την διασύνδεση στην Ευρώπη. Ε, τελευταία ε, πρόσκληση υποβολή προσφορών. Κύριο Σουίτερ, θα του δώσω το λόγο, εφόσον το επιθυμεί. Σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάζετε αυτή την πρόταση υποβολής προσφορών. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διάφορες ε, προτάσεις υποβολής προσφορών για το ΣΕΦ, το Μηχανισμό Διασύνδεσης για την Ευρώπη. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. τα αποτελέσματα της δεύτερης ε, προθεσμίας για το blending call, ε, το, την πρόταση για το ΣΕΖΑΡ είχε την ίδια ημερομηνία καταληκτική. Ε, έχουμε για το 18 προθεσμία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Επίσης έχουμε και το ετήσιο, την ετήσια πρόταση για το 2019 για να ολοκληρώσουμε το project για τον προπολογισμό του ΣΕΦ για την περίοδο αυτή. δύο λόγια για να σας ε, εξηγήσω πώς λειτουργεί το blending. Είναι μια επιχορήγηση που δίδεται. Αυτή τη στιγμή ε, οι δικαιούχοι επιλέγονται και υπογράφουμε την ε, σύμβαση. Οι δικαιούχοι έχουν 12 μήνες για να φτάσουν στην χρηματοδοτική ρήτρα, στο financial close. Έχουν την βεβαιότητα δηλαδή πια ότι θα λάβουν την επιχορήγηση και αυτό θα τους επιτρέψει να διαπραγματευτούν με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το δάνειό τους. Εάν καταφέρουν ε, στη χρηματοδοτική ρήτρα, να φτάσουν στην χρηματοδοτική ρήτρα μέσα στους 12 μήνες, τότε ε, η υπηρεσία η νέα δίνει αυτή την προχρηματοδότηση, την καταβάλει αυτή την προχρηματοδότηση. Επίση, είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα τη πρώτη ανταλλαγή. 39 project ε, ε, εγκρίθηκαν. Ένα δισεκατομμύριο είναι η επιχορήγηση. Όλε οι συμβάσει ε, για την επιχορήγηση έχουν υπογραφεί στο μεταξύ. Και νομίζω δύο από τα έργα έχουν φτάσει ω χρηματοδοτική ρήτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη φάση του blending, της μεικτής αυτής πρότασης, γράφεται στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου για την κινητικότητα, γιατί το δεύτερο πακέτο για την κινητικότητα ε, είχε ένα σχέδιο δράση υπέρ των εναλλακτικών καυσίμων και ο πιο γρήγορος τρόπος για να πλαισιώσουμε ας πούμε, αυτό το δεύτερο πακέτο για την κινητικότητα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ήταν να επεκτείνουμε ε, την προθεσμία της πρότασης ε, προς θέτοντας και ένα προϋπολογισμό 350 εκατομμυρίων ευρώ για τις καινοτόμες και εναλλακτικές πτυχές, εναλλακτικά κάψιμα, καθώς και χρηματοδότηση 115 εκατομμυρίων ευρώ για τα κλασικά έργα. Ως συνήθως, ε, είχαμε πολύ περισσότερες ε, προτάσεις. Ε, ζήτησαν είχαμε με χρηματοδοτήσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Ε, γίνεται μια εξωτερική αξιολόγηση και μειώνει το ποσό αυτό στα 600 εκατομμύρια για ένα προπολογισμό 350 εκατομμύριων όμω συνολικά, έτσι. Έχουμε μια κάποια ευελιξία ε, που περιορίζεται στο 20% και ε, επιλέξαμε κάποια έργα ύψους 404,8 ε, εκατομμύρια ευρώ, που είναι ένα ύψος επενδύσεων 1,8 ε, δισεκατομμύριων ευρώ. Ποια ήταν η προσέγγισή μας για την επιλογή αυτών των έργων. Όπως σας είπα, ο βασικός στόχος αυτής της πρότασης, ε, αυτής της δεύτερης προθεσμής, ήταν να συνοδεύσουμε το σχέδιο δράσης για τα εναλλακτικά καύσιμα ήταν η κόκκινη γραμμή μας σε όλη τη διαδικασία επιλογής. Από 35 επιλεγμένα έργα, τα 26 ε, ανταποκρίνονται σε αυτόν τον ε, προσανατολισμό. Μιλάμε για 23 έργα στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θέλαμε επίσης να εφαρμόσουμε την ίδια αρχή και στους άλλους τομείς. Φερρυπίν, έχουμε δύο έργα στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων της θάλασσας. Ε, που έχουν ε, και αυτά μια, εναλλακτική, μια διάσταση εναλλακτικών καυσίμων, γιατί έχουμε το LNG και CNG, τη διάσταση αυτή, καθώς και ένα έργο σε ένα λιμάνι που έχει ε, τη διάσταση του LNG. πέρα από τα έργα που έχουν σκοπό την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων, έχουμε και ένα χαρτοφυλάκιο έργων πιο κλασικών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των έργων που επιλέξαμε ε, στο πρώτο blending, στην πρώτη προθεσμία του blending και έχουμε ένα σημαντικό έργο στο τομέα των θαλασσίων συνδέσεων. Να σας μιλήσω για κάποια έργα τώρα, έτσι, για να σας παρουσιάσω τη φιλοσοφία. Το σύνολο των έργων που επιλέχθησαν ε, μπορείτε να τα βρείτε στο φυλάδιο που σας μοιράσαμε και υπάρχουν και online. Είναι πληροφορίες βεβαίως που είναι δημόσιες. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι ένα, παράδειγμα, ένα έργο στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας και φυσικού αερίου, ε, συμπιεσμένου φυσικού αερίου, ε, συνδυάζει και τις δύο προσεγγίσεις, δηλαδή μιλάμε για σταθμούς ε, φόρτισης με τέτοιο αέριο και ηλεκτρικούς σταθμούς μεγάλου δυναμικού αλλά και πιο κλασικούς σταθμούς, καθώς και λεωφορεία και αυτοκίνητα σε τέσσερις διαδρόμους. Είναι ένα έργο πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει ολοκληρω... μια ολοκληρωμένη έτσι, φιλοσοφία. Δεν περιορίζεται δηλαδή σε μία μονολύση, αλλά προτείνει μία προσέγγιση πολλαπλή ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα. Ένα έργο λοιπόν που αφορά τέσσερα κρατημέλη για... και μιλάμε για ένα ποσό ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα έργο που αφορά το LNG στον τομέα της θάλασσας όπως ξέρετε έχουμε πολλά έργα σε αυτό το τομέα, γιατί η χρήση του LNG κυρίως για τις θαλάσσιες μεταφορές ε, μικρές, για μικρές και μεσές αποφάσεις, αποστάσεις είναι πολύ σημαντικό για να μειωθεί η τοπική ρήπαση που συνδέεται με τον ντίζελ. Εδώ συνδυάζουμε και τον εξοπλισμό, τον ειδικό για τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και το σταθμό LNG που προβλέπεται στο που είναι πολύτροπο και που επιτρέπει την τροφοδοσία άλλων οχημάτων που χρησιμοποιούμε σε χερσαίες μεταφορές. Είναι ένα έργο, ένα από πολλά τέτοιου είδους και θα κοστίσει 11 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης έχουμε κάποια έργα ε, στον τομέα του υδρογόνου. Επιλέξαμε ένα πολύ σημαντικό ε, στο, στην πρώτη πρόταση υποβολής προσφορών, το πρώτο blending, και τώρα έχουμε και πολλές άλλες προτάσεις τέτοιου τύπου, ε, μιλάμε για χρήση υδρογόνου σε τρεις πόλεις και που συνδυάζει τις υποδομές ε, επαναφόρτησης και καθώς και κινητές μονάδες τροφοδοσίας με υδρογόνου με πολλά λεωφορεία που θα λειτουργούν με υδρογόνο. Ε, πιο πολλές, ε, μιλάμε για πιο μεγάλες επενδύσεις εδώ, 40 εκατομμυρίων ευρώ για, για, μια συνολική επένδυση περίπου μισό δισεκατομμύριο. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τις μεταφορές ε, μεγάλων αποστάσεων εμπορευμάτων με τη χρήση του LNG και εδώ. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι πολύ καινοτόμο γιατί προτείνει όχι μόνο σταθμούς LNG με δύο LNG, αλλά προτείνει και ένα μοντέλο leasing ε, ναύλωσης για τους χρήστες των ε, φορτηγών. γιατί το πρόβλημα εδώ πέρα ε, είναι ότι είναι πολύ πιο ακριβά αυτά τα οχήματα και οι αβεβαιότητες που υπάρχουν ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση τους και την ε, υπολοιπόμενη αξία τους. Εδώ λοιπόν με το leasing, με τη μίσθωση αυτή, μπορούμε να παρακάμψουμε αυτά τα εμπόδια. Και αυτό που προτείνεται είναι ότι οι χρήστες μπορούν να πάρουν το φορτηγό αυτό, να το μισθώσουν δηλαδή, και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους σταθμού τροφοδοσίας του με BOLNG. Μιλάμε για ένα έργο ε, όπου συμμετέχουν έξι κράτη-μέλη, σημαντικός αριθμός, καθώς και επιχειρήσεις στον τομέα των ε, χερσαίων μεταφορών. 25 εκατομμύρια ευρώ ε, επιχορήγηση από τη ΣΕΦ για μια επένδυση ε, ύψους 127 εκατομμύριων ευρώ. Δύο λόγια τώρα για την πρόταση ΣΕΖΑΡ που είχε την ίδια προθεσμία Μιλάμε για μια πρόταση υποβολή προσφορών, ε, όπου ο ενδεικτικό προπολογισμό ήταν 282 ε, εκατομμύρια ευρώ, ε, που είχαμε υπερβολικά πολλές προσφορές και κρατήσαμε στο τέλος τελικά προτάσεις ύψους περίπου ισοδυνάμου με τον προπολογισμό μας. Το μήνυμα το βασικό είναι ότι δώσαμε προτεραιότητα στα έργα τα οποία ε, αφορούν το Caesar Deployment Manager και που έχουν σαν στόχο την ε, δημιουργία αυτού του συστήματος του Caesar. Του Caesar. Τώρα για την πρώτη προβολής προσφορών για το 2018, να σας πω δύο λόγια. Όπως ξέρετε, έχουμε μία πρόταση που τρέχει ακόμα, που είναι πολυετής πρόταση που ξεκίνησε από το 18 από φέτος, ε, ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητων τελειώνει ο ούπο 24 Οκτωβρίου και φέτος αυτή η πρόταση ε, έγινε την ίδια στιγμή με την παρουσίαση του τρίτου πακέτου κινητικότητας, συνέπεσε δηλαδή, και επικεντρώνεται στα θέματα της ψηφιοποίησης, της ασφάλειας στους δρόμους και των πολύτροπων μεταφορών. Ε, προσπαθήσαμε επίσης να συντονίσουμε την παρουσίαση αυτού, αυτής της πρότασης προβολής προσφορών με την πρόταση που αφορά το ΣΕΦ τις, ε, στις τηλεπικοινωνίες, για την κυβερνοασφάλεια, γιατί το θέμα της ε, ψηφιοποίησης στις μεταφορές και της κυβερνοασφάλειας φυσικά συνδέονται άρρηκτα και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να δείξουμε σε επιχειρήσεις και στους φορείς στον τομέα των μεταφορών ότι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ε, στα πλαίσια του ΣΕΦ τηλεπικοινωνίες για το θέμα όμως της κυβερνοασφάλειας. Φτάνουμε λοιπόν στην τελευταία αυτό την πρόσκληση για το 2019 όπως ξέρετε όταν εγκρίθηκε ο παρόν κανονισμός το ΣΕΦ ήθελε το Κοινοβούλιο ένα τμήμα του προϋπολογισμού να διατεθεί στα προγράμματα για το γενικό δίκτυο σφαιρικά και όσον αφορά τα διασυνοριακά τμήματα, υπάρχει ένα ποσοστό για αυτού του είδους επενδύσεις. Στόχος λοιπόν του κόλ του 2019 είναι αυτά τα στοιχεία να καλυφθούν. Είναι για ε, μικρού βεληνικού ε, αυτή η πρόσκληση υποβολή προσφορών με, χαμηλότερα, με χαμηλότερα ποσά, με μείο συνιστώσεις. Ένα τμήμα είναι το διασυνοριακό τμήμα. Εκεί προσθέσαμε και μια συνιστόσα θαλάσσια λιμάνια του δικτύου του γενικού, διότι έτσι διευρύνεται η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν έχουν χερσαίο διασυνολικό τμήμα από το γενικό δίκτυο να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετικές προτάσεις. Και έχουμε μια δεύτερη διάσταση. Πιο μικρή από πλευρά χρημάτων, αλλά πολύ σημαντική. Αφορά τον θόρυβο που προκαλούν οι συνδρομικές μεταφορές. 35 εκατομμύρια ευρώ διαθέσουμε. Έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει δράσεις για το θόρυβο των σιδηροδρόμων και θέλαμε μέσω δράσεων που δρομολογούνται από το 2019 μέχρι το 2022 να μπορέσουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο τμήμα του τροχαίου υλικού για μεταφορά εμπορευμάτων και να παράγουν λιγότερο θόρυβο με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα ανακαίνιση. Από πλευράς διαχείρισης για πρώτη φορά καταφεύγουμε στο unit contribution, συνεισφορά κάθε μονάδας. Μεγάλη απλούστευση για τους δικαιούχους. Δεν έχουν να δικαιολογήσουν το κόστος, πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των βαγονιών που είναι εξοπλισμένα κατάλληλα και με βάση ένα αρχικό τέλος. δεν κάνουμε επαλήθευση του κόστο ε, Εκ των προτέρων καθορίζεται αυτό. Είναι πιο απλά τα πράγματα για του δικαιούχου και αν αυτό είναι επιτυχές είναι μια προσέγγιση που θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε και σε άλλους ε, τομεί. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στην εκτέλεση του προπολογισμού για τις επιχορογήσεις του ΣΕΦ για μεταφορές και αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε συνολικά με αυτά που ανέφερα την πρόσκληση υποβολή ε, ε, προτάσεων το 2018 και 2019, ο συνολικό προπολογισμό για τι επιχορηγήσει διτέθη για τα διάφορα προγράμματα εργασία και 95% ήδη έχει ενταχθεί σε χαρτοφυλάκια επιχορηγήσεων στα πλαίσια των έργων που έχουν δρομολογηθεί και αυτό είναι κάτι που αντιστοιχεί στο 95% του προϋπολογισμού του ΣΕΦ. Και όπως γνωρίζετε, προχωρούμε μέσω ετησίων δόσεων, annual installments. Δεν δεσμεύουμε από πλευρά προπολογισμού το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων, διότι πρόκειται περί ετησίας πρόοδο όσον αφορά τις δεσμεύσεις του προπολογισμού. Είμαστε στο 45% και όσον αφορά τις πληρωμές προχρηματοδότησης ή τελικών ε, οριστικών πληρωμών είμαστε στο 20% του προγραμματισμού. Άρα, κλείνοντας, λέγω ότι βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως και αναφέρθηκε, να έχουμε και άλλες ε, προσκλήσεις υποβολή ε, προσφορών. Αυτές οι διαδικασίες θα ενταχθούν στο νέο προγραμματισμό Use it or lose it. Αυτό θα ξεκινήσει από αρχές του επόμενου έτους. Για να έχουμε και υποβολές προσφορών για το 2020 για βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αυτού του τομέα του ΣΕΦ. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσουμε το λόγο στα μέλη μας. Ο κ. Βιμ Βάντερκαμπ. Πρόεδρε, μήπως είναι δυνατόν να δούμε εδώ τη διαφάνεια για το 2018, την πρόσθεση δηλαδή υποβολή προτάσεων του 2018. Γιατί δεν κατάλαβα αν τελικά περιλαμβάνεται κανονικά ε, έργα ή όχι. Deze, ja, dank u. Ναι, αυτή τη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι εξή. Έχουμε να κάνουμε μόνο με την ψηφιοποίηση των ζητημάτων ασφαλεία στις οδικέ μεταφορά και την πολυτροπικότητα των μεταφορών. Άρα λοιπόν άλλο, άλλα έργα διαφορετικά, δηλαδή διαφορετική φύση, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη εδώ, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Τώρα, στην δεύτερη, ή μάλλον στην τελευταία διαφάνεια, ξεκινάμε με αυτήν την λογική του use it or lose it. Δηλαδή αξιοποίηση των κοντιλίων. Ε, μη αξιοποίησή τους. Ε, είδαμε για παράδειγμα εδώ καταβολή του 20%. Άρα λοιπόν από πότε ξεκινάει αυτή η συλλογιστική ε, του Use it or lose it από το 2020, από το 2029. Πότε λοιπόν αρχίζει να ισχύει αυτό το σύστημα, δηλαδή το αξιοποιεί κανείς τα κονδύλια ή τα χάνει. Και από την άλλη μεριά είχαμε ε, μία κανονική πρόσκληση υποβολή σε προτάσεων 350 δισεκατομμυρίων ε, συμπληρωματικά προ εκείνο των 2 δισεκατομμυρίων. Δεν, κα, δεν κατάλαβα κάτι. Δηλαδή υπάρχει μία δεύτερη πρόσκληση υποβολή προτάσεων για κανονικά project. σω εγώ να μην κατάλαβα κάτι. Ευχαριστώ. Και φυσικά σε ευχαριστώ και για αυτή την παρουσίαση. Μετά με κυρία Γιάλα Σέντορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε σε κάποια προγράμματα βλέπω ότι εντοπίζονται σαν διάδρομοι βόρειο Μεσογειακή κλπ. Αλλά στη Βόρεια Θάλασσα. Λοιπόν, όταν είδα, είδα και για τις νότιες θάλασσες. Ουσιαστικά οι διάδρομοι αυτοί που αναφέρονται αφορούν τη Βόρεια Θάλασσα. Μιλάμε για διαδρόμους του Βορρά ή μεταξύ Λονδίνου, Κοπενχάγης, Ρήγας. Ελάχιστα αναφέρω τη Μεσόγειος στη γεωγραφική προσέγγιση. Μου φαίνεται κάτι αντιφατικό. Εκφράζουμε ικανοποίηση αρχικά ότι κάτι έγινε τη Μεσόγειο και όταν εξετάζουμε προσεκτικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει τίποτα για τη Μεσόγειο. Για πολλά προγράμματα είναι για να πληρωθούν λεωφορεία, φορτηγά και αυτοκίνητα στο Παρίσι κλπ. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Το πρόγραμμα τι χρηματοδοτεί πέρα από τους σταθμούς και τα αυτοκίνητα και τα οχήματα, τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από τις εξηγήσει. Λίγε διευκρινήσει θα ήθελα από αυτού. Τι ακριβώς χρηματοδοτείται σε κάποιες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι ίσως οι εξηγήσει δεν είναι σαφείς. Όσον αφορά τους δικαιούχους, είναι δυνατόν να αγοράσει και να αγοράσει ολόκληρους στόλους αυτοκινήτων, λεωφορείων. Μήπως μπορείτε να το εξηγήσετε καλύτερα για να ξέρουμε τι ακριβώς χρηματοδοτούμε. Διότι έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε γρήγορα ε, τη μείωση της αστικής ε, ρήπανσης. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεμόντε, όχι. Κοιτάξτε, φιλομέτρησα την έκθεση. Πολύ, αντίθετα, εγώ θα έλεγα ότι υπήρχαν προλά προγράμματα του Νότου. Πολύ Ισπανία είδα εγώ. Διάλογος εκτός μικροφώνου. Βλέπω ότι Ρένφε, Βαρκελόνη, Πέρτο Σέντρο, Βαρκελόνη, Ραβένα. Πάντα στο Νότο βρισκόμαστε. Λοιπόν, κάποιες απαντήσεις ίσως να μας δώσει. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την υποβολή προσφορών του προτάσεων του 2018, είμαστε στο τέλος του προϋπολογισμού και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε, να προκηρύξουμε πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Είπαμε να εστιαστούμε επί περιορισμένων θεμάτων και γι' αυτό έχουμε θεματική προσέγγιση, ψηφιοποίηση, οδική ασφάλεια και πολυτροπικότητα. Δεν υπήρξε γενική ε, πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Όσον αφορά την αρχή «use it or lose it», δεν είναι ότι ξεκινά για όλα τα προγράμματα συγκεκριμένη ημερομηνία, εξαρτάται από το κάθε έργο από τη Συμφωνία Επιχορήγησης. Κάποια προγράμματα έληξαν φέτος, Φερρυπίν, Δεκέμβρη του 2018, λίγουν μάλλον, και σε κάποιες περιπτώσεις εγκρίναμε ε, παράταση λόγω καθυστέρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν ξεκίνησαν καθόλου τα έργα, ακόμα και με παράταση δεν θα μπορούσαν να μας εγγυηθούν ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν το έργο. Εν αυτή η περιπτώση προτιμήσαμε να πούμε συγγνώμη, είχατε την ευκαιρία σας, δεν εγκρίνουμε παράταση και αυτό σημαίνει ότι το ποσό που ήταν στη συμφωνία επιχορήγησης εν μέρη συνολικά επιστρέψει στο Ταμείο και θα ξαναχρησιμοποιηθεί για τον επόμενο κύκλο υποβολή προσφορών. Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία υποβολή προτάσεων χρειάζεται μια, κριτική, ε, μια κρίσιμη μάζα. Και γι' αυτό κάνουν τη διαδικασία σε τμήματα. Όλες τις συμφωνίες εξετάσαμε φέτος που εξέπνεαν από τώρα μέχρι άνοιξη του 19 διότι έπρεπε γρήγορα να πάρουμε απόφαση αν θα σταματήσουμε, θα παρατείνουμε, τι θα κάνουμε με όλους αυτούς. Και για τα υπόλοιπα που έχουν έναν ορίζοντα λήξεως το 2020 ή 2021 θα πρέπει να αποφασίσουμε αρχές του 19 για να αλλάξουμε τη συμφωνία των υποχρεωγήσεων Άνοιξη του 19 είναι η καλή στιγμή. Εάν κάνουμε αλλαγέ στην άνοιξη του 2019, μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα το αργότερο τέλο 19 και ξανά να κάνουμε διαδικασία υποβολή προσφορών που να, είναι χρήσιμη. Διότι η επιστροφή χρημάτων και η πρόσκληση υποβολή προτάσεων είναι κάτι, αλλά χρειάζεται και επαρκή περίοδο υλοποίηση των έργων. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το τέλο του 2023. Αν θέλουμε να έχουμε μια χρήσιμη διαδικασία επανάκτηση χρημάτων, δεν μπορεί να ξεκινήσει προς το τέλος των προγραμμάτων. Το 2020 είναι η σωστή χρονιά, ίσως τελευταία χρονιά για τις μεγάλες διαδικασίες υποβολής προσφορών και αν έχουμε πολλές προσφορές θα πρέπει το 2020 να μπορούμε να ξεκινήσουμε άρα και να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες που έχουμε κάνει μέχρι το 2019 για τις επιχορηγήσεις. Όσον αφορά τα κινητά στοιχεία περιουσίας αν θέλετε, στόλους οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, δεν τα χρηματοδοτούμε έτσι γενικά. Πολλά προγράμματα συμπεριλαμβάνουν στόλους, λεωφορείων κλπ. Αυτό που χρηματοδοτούμε είναι η διαφορά μεταξύ κανονικού διζελοκίνητου λεωφορείου και λεωφορείου με υγροποιημένο φυσικό αέριο ή με υδρογόνο. Χρηματοδοτούμε τη διαφορά. Αυτή είναι η βάση κόστος και από εκεί χρηματοδοτούμε το 20% ελάχιστο ποσοστό αυτού που χρηματοδοτούμε από τα ε, κινητά στοιχεία ενεργητικού. Εντός, εκτός, ο διάλογος εκτός μικροφών. 20% της διαφοράς του κόστους. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά είναι ένα μήνυμα που δίνουμε και αυτού του είδους τα προγράμματα. Εν γέννη χρηματοδοτούμε κυρίως υποδομές για τα κάψιμα Φερρυπίν η τροφοδότηση καύσιμα. Εδώ χρηματοδοτούμε τη διαφορά κόστους εν μέρη ή συνολικά για την αλλαγή τεχνολογίας στο στόλο. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι έχουμε βάλει ανώτατο όριο όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση της διαφοράς. Διότι έχουμε στοιχεία από την αγορά και δεν έχουμε χρηματοδοτήσει αυτό που ζητούσε ο δικαιούχος αλλά θέσαμε ένα ανώτατο όριο σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο. Αυτά και ευχαριστώ. Ο κ. Καμπ παλι πάλι. Έχω κάποιες ερωτήσεις, μία-δύο ερωτήσεις και έχουμε και κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας. Η πρώτη ερώτηση. Μας δείξατε τα στοιχεία για αυτή την ανάμειξη, για το blending. Ένα στοιχείο ένα δισεκατομμύριο ευρώ και μετά 350 εκατομμύρια και μετά έχετε και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από αυτή την ανάμειξη από το blending. Ποια είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όλα αυτά. Τα υπόλοιπα των χρημάτων από την ΕΚΤ έρχονται από δημόσιες τράπεζες, προέρχονται από κρατικές τράπεζες. Τα υπόλοιπα χρήματα από πού προέρχονται. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Στον Ολλανδικό τύπο, εδώ και 15 μέρες, διαβάσαμε μία έκθεση. Με ένα δημοσίευμα. Α, ναι, ναι, ναι. Είπατε, Ευρω... είπα ΕΚΤ, όχι, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εννοούσα, όχι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ο Βαντεν Κάμπ». Μιλούσε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η δεύτερη ερώτηση, λοιπόν. Στον τύπο, τον Ολλανδικό, εδώ και 15 μέρες, υπήρχε ένα άρθρο και έλεγε ότι 273 εκατομμύρια από το τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, κυρίως από τις χώρες συνοχής κάποια από αυτά τα χρήματα μπαίνουν στο ΣΕΦ ή το ΣΕΦ είναι εντελώ διαφοροποιημένο από αυτό το στοιχείο που παρουσιάστηκε στον Ολλανδικό τύπο. Είναι η ερώτηση. Η απάντηση. Ευχαριστώ. Για το προπολογισμό. Αρχικά είχαμε ένα δις για το πρώτο building, ε, blending πέρσι. 39 προγράμματα εγκρίθηκαν, συμφωνίες υπεγράφησαν. Όταν παρουσιάσαμε το δεύτερο πακέτο κινητικότητας, θέλαμε να το συνοδεύσουμε με κάποια οικονομική υποστήριξη. Ταχύτερος τρόπος ήταν να κρατήσουμε ανοιχτό το διαγωνισμό υποβολή προσφορών με το blending με δεύτερη προθεσμία και να δώσουμε και άλλα 350 εκατομμύρια. Επειδή έχουμε κάποια ευελιξία, πήγαμε λίγο πιο πάνω από τα 350. Το συνολικό πρόγραμμα για το blending 1 και 2 είναι ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια. Μετά, ποια είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι ανοιχτό το πεδίο. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι εταίρος για κάποια προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με το Ταμείο Εγγύσεων του ΕΦΣΥ, αλλά το τεράστιο ποσοστό από τα προγράμματα δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά από διάφορες εθνικές εμπορικές τράπεζες. Οπότε τα αφήσαμε ανοιχτό. Ο δικαιούχο επιλέγει τον ε, εταίρο, τον χρηματοδοτικό εταίρο που προτιμάει. Δεύτερη ερώτηση. Τα χρήματα που δεν δαπανήθηκαν, που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ναι, απάντηση δεν σχετίζεται με το ΣΕΦ. 100% διατίθεται. Δεν υπάρχουν χρήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Βαντεγκάμπ. Καλώς. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για την παρουσίασή σας, για τη θεσιμότητά σας. Λοιπόν, τελειώσαμε πιο νωρί. Ευχαριστώ του γενναίου που ήταν παρόντε. Ευχαριστούμε και του διερμηνεί που και μια φορά τελείωσαν ε, πιο νωρί που δεν είναι και πολύ συχνό φαινόμενο. Ευχαριστώ όλους. Επόμενη συνεδρίαση στις 5 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Θα επανέλθει ο πρόεδρος τότε.